Mes chers collègues, nous Συνεχίζουμε. Υποδέχομαι τον κύριο Μίλη, Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Θαλάσσια Ασφάλεια. Τον ευχαριστώ για τις τακτικές επισκέψεις του κατά τη διάρκεια της εντολής σας Οργανώσατε επίσης και τις νέες ε, αρμοδιότητές σας, όπως το νέο πρόγραμμα για τη Μεσόγειο, το θέμα της ε, θαλάσσιας μόλυνσης από τις ε, θαλάσσιες πλατφόρμες εξόριξης πετρελαίου, όπως επίσης και τη νέα συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών θείου. Όλα αυτά Είναι ιδιαίτερο ενδιαφέροντα να υπογραμμίσω επίσης και τον σημαντικό ρόλο της υπηρεσίας σας στον τομέα του ελέγχου των σκαφών, έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των σκαφών που δεν είναι σύμβατα με θέματα, σε θέματα ασφάλειας και σε επίπεδο επίσης οικολογικό, δηλαδή τα πράγματα εξαρτώνται κατά πολύ τελικά από τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε. Έχετε επανειλημμένα ζητήσει την ενίσχυση των οικονομικών μέσων, τα οποία έχει η ΕΜΣΑ στη διάθεσή της, για να φέρετε εις πέρα στην αποστολή την οποία έχετε αναλάβει. Είμαι πάντως πεπισμένη ότι εμείς θα συνεχίσουμε να σας συνδράμουμε και θα ήθελα να συζητήσω να μας παρουσιάσετε τις δραστηριότητές σας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους έτσι ώστε να δούμε και ποιες θα είναι οι φετινές προκλήσεις. Μετά την παρουσίασή σας θα ξεκινήσει η συζήτηση με τους αγαπητούς συναδέλφους. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Για μια ακόμη φορά θέλω να σας συγχαρώ για το διορισμό σας στην θέση της Προέδρου αυτής της σημαντικής επιτροπής για μας. Κυρίες και κύριοι, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την Επιτροπή σας γιατί μου δώσατε τη δυνατότητα να σας ενημερώσω για τις δραστηριότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΜΣΑ είναι σημαντικό για μένα και για το προσωπικό της ΕΜΣΑ το ότι σε αιτήσια βάση μπορούμε να σας παρουσιάζουμε τις προτεραιότητές μας για τους επόμενους μήνες. Βασικό στόχος της ΕΜΣΑ για το 2017 είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις ε, κομβικές, τις κεντρικές υπηρεσίες με τα αδιαθέσιμα μέσα ε, σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Η υποστήριξή σας επαληθεύθηκε και τον προηγούμενο Οκτώβριο με την τελευταία τροπολόγηση στον ιδρυτικό μας κανονισμό που καθιστά την υπηρεσία μας κομβικό παίκτη σε σχέση με την ακτοφυλακή πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προσπάθειές μας για να φτάσουμε στην κορυφή του προσωπικού που χρειαζόμαστε θα συνεχιστεί το 2017. Συνολικά στο τέλος του χρόνου θα έχουμε πετύχει 10% μείωση. Παράλληλα, όπως βλέπετε στο γράφημα αυτό, η διευρυμένη αποστολή μας, η διευρυμένη αρμοδιότητά μας συνοδεύτηκε και από νέους πόρους έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της συμμετοχής μας στην ακτοφυλακή. Η στήριξη της αποστολής σε επίπεδο ακτοφυλακής δεν είναι κάτι το, το καινούριο για μας. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί εδώ και καιρό σαν τμήμα των επιθεωρήσεων της όσες κάνουμε. Αυτό το οποίο αλλάζει τώρα είναι πραγματικά το μέγεθος, το μεγάλο μέγεθος αυτής της αποστολής, αυτού του ρόλου όπως επίσης και ο αριθμός των τοπικών αρχών που θα αποφεληθούν από την δραστηριότητά μας. Το 2017 λοιπόν θα συνεργαστούμε με την ΕΦΚΑ και το Frontex σε τρεις τομείς, καταρχάς συλλογή δεδομένων, βελτίωση των δυνατοτήτων με νέες τεχνολογίες και νέες δραστηριότητες αύξησης της ικανότητάς μας, των ικανοτήτων μας. Σήμερα η είναι αν θέλετε η βασική εικόνα, παρέχει τη βασική εικόνα της ε, ναυσιπλοείας στην Ευρώπη. 19 ε, εκατομμύρια μηνύματα και στοιχεία την ημέρα ανταλλάσσονται με βάση τα συστήματά μας ανάμεσα στα σκάφη και τις ε, υπηρεσίες εδάφους. Αυτή η εικόνα είναι φυσικά διαθέσιμη στις εθνικές και τοπικές αρχές για διάφορους λόγους και υποστηρίζοντας τις διάφορες αποστολές γύρω από την ακτοφυλακή με βάση την κατανομή των αρμοδιοτήτων. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την ΕΦΚΑ και το Frontex για να έχουμε πάντα μια πλήρη και ακριβή εικόνα. Οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε σε πραγματικό χρόνο είναι απαραίτητες έτσι ώστε να λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις οι οποίες ε, πληροφορίες και στοιχεία είναι πλέον διαθέσιμες και σε φορητά μέσα όπως ε, τα έξυπνα τηλέφωνα, τα ευφυή τηλέφωνα. Οι τεχνολογίες εξελίσσονται με μεγάλη ταχύτητα. Η ΕΜΣΑ, σύμφωνα και με το πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει, προσπάθησε το 2016 να διασφαλίσει αρκετές υπηρεσίες και μέσω μη επανδρομένων αεροσκαφών. Σύντομα θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε νέες υπηρεσίες προς τις τοπικές αρχές, ε, υποστηρίζοντας πάρα πολλές δραστηριότητες γύρω από την βασική αποστολή που είναι η ακτοφυλακή. τα μη επανδρομένα αυτά είτε ε, τύπου ελικοπτέρων είτε τύπου αεροσκαφών θα είναι διαθέσιμα για υπηρεσίες όπως ο έλεγχος των συνόρων, η ασφάλεια της ε, ναυσιπλοείας, έρευνα και διάσωση, ε, επιβολή του νόμου κτλ. η ενίσχυση των αποστολών μας στον τομέα της ακτοφυλακής σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να αποκτήσουμε ικανότητες και να καταρτιστούμε αντίστοιχα. Χρησιμοποιούμε ε, διάφορα συστήματα εκμάθησης των αποστολών μας σε επίπεδο σαν παράδειγμα φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων αυτά τα συστήματα τα οποία είναι διαθέσιμα σε επίπεδο λογισμικού θα χρησιμοποιηθούν για την διεύρυνση και την εμβάθυνση των ικανοτήτων σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε 18 διδακτικά τέτοια συστήματα για θέματα διαφορετικά μεταξύ τους όπως η ασφάλεια, η στίβαξη των εμπορευμάτων κτλ. Δημοσιεύουμε επίσης μια ετήσια έκθεση για τα θύματα στις θαλάσσιες μεταφορές και για τα ατυχήματα και το κάναμε και για το 2016. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται συνεχώς από ό,τι δείχνουν οι στατιστικές οι οποίες γίνονται σε ετήσια βάση πιο αντιπροσωπευτικές. Η καινοτομία από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο είναι η δημοσίευση στοιχείων για τη διερεύνηση ατυχημάτων ε, σε ε, τριμηνιαία βάση, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει καλύτερη πρόληψη. Οι στατιστικές τις οποίες έχουμε για το προσωπικό των σκαφών, τους ναυτεργάτες, έχουμε συγκεκριμένους αριθμούς για αυτούς οι οποίοι εργάζονται έχοντας συγκεκριμένα πιστοποιητικά και είναι ο πρώτος χρόνος που έχουμε πλήρη στοιχεία. Θα συνεχίσουμε να συλλέγουμε τα στοιχεία τους επόμενους χρόνους και έτσι θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα την φύση του εργατικού δυναμικού στον τομέα της ναυτιλίας. Θα συνεχίσουμε εμείς να εκτείνουμε και την εμβέλεια του συστήματος θέτης. Το σύστημα αυτό υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε ε, κυρίως στην αρχή για λιμενικούς ελέγχους, αλλά θα καλύψει και ε, άλλα θέματα ελέγχους και επιθεωρήσεις που προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο. Σαν παράδειγμα... Ε, January 2015 to record information related to the implementation of the revised sulfur directive. Ε, σύμφωνα με την οδηγία για το θείο, σαν παράδειγμα οι έλεγχοι που κάνουμε δίδουν ήδη εξαιρετικά αποτελέσματα. Επίσης θα εξελίξουμε και το σύστημα MRV για τις εκπομπές διοξιδίου άνθρακα από τους στόλους. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αποστολή και πρόκληση για μας. Θα είναι το πρώτο σύστημα διαθέσιμο και ικανό να διαδράσει όχι μόνο με τα εθνικά στοιχεία, αλλά και τις επιχειρήσεις στον υπόλοιπο κόσμο. Την Άνοιξη θα ξεκινήσουμε ε, μια νέα σειρά προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ε, για τη Μεσόγειο, την Κασπία και τη Μαύρη Θάλασσα. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στην πολιτική της Ένωσης απέναντι στις χώρες, της παράκτιες αυτών των περιοχών ε, και σκοπεύει στην επιβολή κανόνων και ρυθμίσεων αντιστοίχων με αυτές που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια πρώτα βήματα έχουν γίνει με επιτυχία ε, με τα δίκτυα στα οποία έχει ήδη υπάρξει έλεγχος στις γειτονικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιοχές. Ε, σχετικά τώρα με τη διευκόλυνση της, των θαλασσίων μεταφορών, εμείς υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έμεσα και την ε, βιομηχανία την ναυτιλιακή σε σχέση με τους ελέγχους στους λιμένες. Αποτελούμε τμήμα ενός πιλωτικού προγράμματος το οποίο θα οδηγήσει στο πρωτότυπο της ενιαίας θηρίδας καταγραφής κινήσεων στον τομέα της ναυτιλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα πολύ σημαντικό ε, θέμα είναι η διασφάλιση ε, στοιχείων γεωεντοπισμού δορυφορικού τύπου στην ουσία θα επικυρώνουμε ε, στοιχεία τα οποία θα δημιουργούν περισσότερη βεβαιότητα για τον γεωεντοπισμό των σκαφών. Ε, αυτά τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα για τα σκάφη όταν ε, πλέουν μακράν των ακτών. Είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για πλοία τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο, όταν βρίσκονται εκτός των χωρικών υδάτων, και τα δορυφορικά αυτά στοιχεία μερικές φορές θα είναι και τα μοναδικά ικανά να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε το σκάφος. Ήδη από το προηγούμενο φθινόπωρο εμείς ε, υπογράψαμε ένα συμβόλαιο έτσι ώστε να τροφοδοτούμε το σύστημα αυτό με δορυφορικού τύπου στα στοιχεία. Το Κοπέρνικους είναι το δορυφορικό πρόγραμμα παρακολούθησης ε, της επιφάνειας της γης και χρησιμοποιείται και για τον έλεγχο της ναυσιπλοείας. Νομίζω ότι λίγους μήνες μετά την θέση σε λειτουργία του συστήματος Κοπέρνικους έχει ήδη αποδείξει την προστιθέμενη αξία την οποία μπορεί να παρέχει αυξάνοντας ε, ε, την ασφάλεια, καταπολεμώντας το λαθρεμπόριο ναρκωτικών κτλ οι υπηρεσίες γύρω από το Κοπέρνητους ε, θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο για την έβρεση, σαν παράδειγμα ανείχνευση και έβρεση εμπορευματοκιβωτίων τα οποία έχουν πέσει στη θάλασσα. Και ταυτόχρονα θα βοηθήσουμε και για την καταπολέμηση της μόλυνσης στις παράκτιες περιοχές. Έχουμε οκτώ σκάφη τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία Όλα αυτά τα σημεία, ε, όλα αυτά τα σκάφη λειτουργούν μέσω της συνεργασίας του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα και ε, παρέχουμε τα μέσα εξοπλισμού τους. Αλλά τα μέσα αυτά τα λειτουργούν ιδιωτικές εταιρείες με ε, ναυτικούς οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και οι οποίοι έχουν υπογράψει συμβάσεις stand-by με την ΕΜΣΑ για παρέμβαση μέσα σε 24 ώρες όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Προσπαθούμε επίσης ε, να πλουτίζουμε τον εξοπλισμό μας για την καταπολέμηση της μόλυνσης από πετρέλαιο, δημιουργώντας ένα δίκτυο <coughs> συμπληρωματικό με τα σκάφη τα οποία προανέφερα, χρησιμοποιούμε μέσα τα οποία είναι μέσα αποκλεισμού περιοχών ναυτικών και δεν είναι διαθέσιμα σε άλλες υπηρεσίες εκτός από τις ειδικέ μας και θα ξεκινήσουν να ισχύουν και για περιοχές όπως η Αδριατική. Ελπίζω ότι αυτή η επιλεκτική, αν θέλετε, περιγραφή των προτεραιοτήτων μας για το 2017 να σας έχουν δώσει ένα μικρό μόνο τμήμα των δραστηριοτήτων μας. Έχετε μία μόνιμη πρόσκληση για να επισκεφθείτε την έμσα στην πόλη της Λισαβόνας και η επίσκεψη τον προηγούμενο Μάρτιο, Μάρτιο συγγνώμη, της κυρίας Μοντέιρο Αγουιλάρη ήταν ιδιαίτερος ενδιαφέρουσα. Euh, euh, euh, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε για την πραγματικά ευρία και πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση των δραστηριοτήτων σας. Ας αρχίσουμε τώρα την συζήτηση με τους συντονιστές και πρώτος ο κύριος Βάντιν Κάμπ. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που είναι εδώ και η Κλάντια Μοντέρο και ελπίζω μετά από μένα να έχει και αυτή την ευκαιρία να θέσει ορισμένα ερωτήματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή για την παρουσίασή του. Εάν κατάλαβα καλά, εξελίσσεστε από μια κλασική υπηρεσία ασφαλείας σε μία υπηρεσία, σε έναν φορέα που θα ασχολείται περισσότερο με την διαφύλαξη ε, των παράκτων περιοχών, τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και με την καινοτομία. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα δορυφορικά και το Κοπέρνικο. Πώς τα κάνετε όλα αυτά. Θεωρώ εξαιρετικά θετική την εξέλιξη αυτή. Όμως έχετε το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, τους απαραίτητους πόρους. Ξέρετε ότι εμείς ως ε, πολιτικοί ποτέ δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ό,τι και να κάνετε καλά, εμείς θα σας λέμε τι μπορείτε να κάνετε ακόμα καλύτερα. Και ανεβάζουμε και άλλο τον πύχη. Έτσι θα ήθελα να σας ρωτήσω, μέχρι πού φτάνετε στη Μεσόγειο. Περιορίζετε στα χωρικά ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι το ρωτώ αυτό σε σχέση με αυτά τα σκάφη, τις βάρκες μάλλον, ε, με τις οποίες ταξιδεύουν οι αιτούντες άσυλο. Ε, κάποιο ρόλο, ενδεχομένως αποτρεπτικό, για να μην ξεκινούν αυτές οι βάρκες από ε, τις νότιες ακτές της Μεσογείου. Έχετε λοιπόν μια τέτοια ιδιότητα οργανισμού ασφαλείας και μετά γνωρίζετε τι κάνουν οι υπόλοιπε υπηρεσίε ή μία, ποιες είναι οι αρμοδιότητε της άλλη. και αυτό ήθελα να το θίξω. Μετά, σε ό,τι αφορά ε, και στην Επιτροπή ΕΝΒΗ έχουν συζητήθει τα ζητήματα του IMO και του ΕΦΣΙ και χαίρομαι που τα αναφέρατε κι εσείς, όμως ε, δεν ξέρω κατά πόσο Μπορεί να υπάρξει μια ευρωπαϊκή ε, προοπτική για το ETS και αν αυτό είναι ε, σκόπιμη επιλογή. Είναι πολιτικό βέβαια το ζήτημα, αλλά ήθελα να το θίξω. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παντρικάμπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και για αυτή τη δυνατότητα που μου δίνετε ε, να πάρω το λόγο και να σας συγχαρώ για την εκλογή σας. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μίλη της ΕΜΣΑ, παρακολουθήσαμε τη συζήτηση και με τους άλλους συναδέλφους και γνωρίζουμε ποια είναι η προϊστορία της συγκεκριμένης υπηρεσίας και την ανάγκη η οποία υπάρχει να καλυφθούν όλα αυτά τα μέτωπα και όχι μόνο λίγα από αυτά όπως το θέμα του εντοπισμού των σκαφών. Τώρα λοιπόν η ΕΜΣΑ έχει αρκετά μέσα έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά της, αλλά όπως είπε και ο κύριος Βαντερκάμπ ε, μπαίνει πλέον και σε άλλα χωράφια τα οποία είναι πιο περίπλοκα, σε άλλα πλαίσια, αλλά νομίζω ότι η αρχική εντολή η οποία ήταν να διασφαλίσει τον έλεγχο των θαλασσίων μεταφορών, ο οποίος μετά από την κρίση, ε, από διάφορες κρίσεις κατάφερε να αναγεννηθεί. και να καλύψει τομείς όπως και η προστασία του, ε, των θαλασσίων περιοχών πέρα από τις δραστηριότητες τις παραδοσιακές όπως είναι τα θέματα ασφάλειας. Ο, για όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν οι εγγύησει που απαιτούνται μέσω της νέας εντολής και σε συνεργασία με την Frontex καλείται να διαχειριστεί όλο και πιο ε, περισσότερο μάλλον περίπλοκες καταστάσεις και αυτό μάλιστα και με ε, ουσιαστικά μειούμενους ανθρώπινους πόρους γενικότερα και η κατάσταση θα πρέπει να βελτιωθεί γιατί εμείς θέλουμε να υπάρξει ένα βήμα θετικό και μια αναπτυξιακή ε, τάση και γι' αυτό ακριβώς ε, θεωρούμε ότι και για τη δική μας χώρα η προσπάθεια σας είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σέντερ. Ο επόμενος, Ζέλα. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που βλέπουμε εδώ το Γενικό Διευθυντή. Πάντα κάνατε μια πολύ καλή παρουσίαση. Θα ήθελα να θέσω τα εξή δύο ερωτήματα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τις νέες αρμοδιότητες με την ε, ακτοφυλακή και το θέμα το μεταναστευτικό. Πριν από 1,5 χρόνο επισκεφθήκαμε τη Λισαβόνα μόλις ξεκινούσατε δεν είχατε τους πόρους. Τώρα από ό,τι κατάλαβα έχετε 15 υπαλλήλου. Μπορείτε να μας δώσετε απλά παραδείγματα των νέων αρμοδιοτήτων σας. Γιατί από τα μέσα ενημέρωσης αναφέρεται ότι το πρόβλημα δεν είναι ο εντοπισμός ε, των ε, διακινητών. Το θέμα είναι ότι πριν την αναχώρηση των ε, σκαφών αυτών ε, υπάρχουν ακόμα και μη κυβερνητικέ οργανώσεις που εμπλέκονται σε αυτό και μπορούν να φύγουν ε, σε μία ακτίνα έως 20 ναυτικά μίλια. Αυτό είναι το πρώτο λοιπόν. Το δεύτερο, αρκετά αφελές, ρώτησα σήμερα το πρωί και τη Μαλτέζικη Προεδρία και δεν πήρα απάντηση. Στη Βόρεια Θάλασσα και στην Βαλτική Θάλασσα έχουν αλλάξει από το 2015 οι εκπομπές ε, αερίων του θερμοκηπίου. Ξέρω ότι είναι λεπτό το ζήτημα, αλλά δεν έχει έρθει η ώρα να αρχίσουμε να εξετάζουμε και για τη Μεσόγειο. Τι συμβαίνει. Να θίξουμε και το ίδιο ζήτημα και εκεί, γιατί πρόκειται για ρήπατσα και πάλι. Και βεβαίω η Μεσόγειος έχει πολύ ψηλή κίνηση. Ευχαριστούμε. Κύριε Τιτίνκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Στελίτσκα, καλώς ήρθατε κύριε Γενική Διευθυντά. Κάποιες ερωτήσεις έχουν ήδη διτεθεί από τους συναδέλφους. Θα είμαι λοιπόν ε, σύντομος. Στην παρουσίασή σας, παρότι ήταν πολύ περίπλογη και εμπεριστατωμένη, ε, έλειπε κάτι, κατά τη γνώμη μου. Τι δεν πάει καλά που υπάρχουν αδυναμίες, ελλείψεις ως προς τις ε, φιλοδοξίες μας και τα χρονοδιαγράμματά μας. Και σε... είναι η στενοπή που αντιμετωπίζουμε. Κατάλαβε από αυτά που είπατε ότι είναι πολύ υψηλέ αρμοδιότητε και απαιτητικέ, όμω εμεί πώ μπορούμε να σα βοηθήσουμε. Τι σας παρουσιάζει δυσκολία. Δεύτερον, πολύ χαίρομαι που μας δώσατε και την ε, παρουσίαση αυτή για την αλληλεπίδραση με τον Κοπέρνικο. Όμως ε, και πάλι να έχετε κατά νου ότι σε πολλούς άλλους τομείς ε, απέχουμε πολύ από το να αξιοποιήσουμε τα όσα μας παρέχουν ο Γαλιλαίος και ο Κοπέρνικος. Τι θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να διερευνήσουμε περαιτέρω και κατά κάποιον τρόπο καθυστερούμε. γιατί πραγματικά έχω την αίσθηση ότι οι ευκαιρίες που προσφέρονται είναι πολύ ψηλότερες σε σχέση με την, ε, για την παροχή υπηρεσίων σε σχέση με αυτά που καταφέρνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τέιλορ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας βλέπω και πάλι, κύριε Μουλή. Νομίζω όλοι οι υπόλοιποι θέτουν τα ίδια ερωτήματα. Το ίδιο ερώτημα θα το θέσω και εγώ για λόγους αφήνειας. Με έχει εντυπωσιάσει το έργο της ΕΜΣΑ με την πάρτα των ετών. Πέρυσι σας δώσαμε επιπλέον αρμοδιότητα και καθήκον να παρακολουθείτε και την, ε, τις υποδομές ε, εξόριξης ε, πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και τη συνδρομή στη Frontex για την ακτοφυλακή. Και μαζί με όλους τους υπόλοιπους μπορώ και εγώ να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι υπάρχουν αναδυόμενες πιέσεις σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων σας και την επιτέλεση των καθηκόντων σας. Ευχαριστούμε κύριε Τέιλερ. Κυρία Κιλόνεν. Με το που ήρθατε, σας δίνουμε και το λόγο κατευθείαν. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για το προσφυγικό ζήτημα. το οποίο δεν θίγεται τόσο πολύ. Όμως, από τον κλάδο των ε, θαλάσσιων μεταφορών, κατανοώ ότι δεν έχει επιληθεί το πρόβλημα. Τι νομίζετε ότι θα πρέπει να κάνει το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την κατάσταση των προσφύγων σε σύνδεση και με την ε, ασφάλεια στη θάλασσα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Φώστερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Μερικές παρατηρήσεις μόνο, γιατί κάποιες άλλες έχουν καλυφθεί από τους συναδέλφους. Κατά την ε, ε, εισαγωγή της οδηγίας για το θείο υπήρχε ένα θέμα. Υπήρχαν πολλές προκλήσεις για την ίδια την αυσιπλοεία σε ό,τι αφορά την επικαιροποίηση ε, της τεχνολογίας. Και ξέρετε ότι είναι μια εξαιρετικά ταπανηρή διαδικασία. Πέραν τούτου, ανεξάρτητα από το κατά πόσο αυτό αφορά μόνο τη Βόρεια Θάλασσα ή και τη Μεσόγειο, είχαμε ένα ζήτημα πέρσι και το είχαμε θίξει. Είχαμε λοιπόν σκάφη που, ε, στα οποία είχε κατασταθεί όλο, όλη η καινούργια τεχνολογία και ο εξοπλισμός και σε ορισμένους ε, λιμένες ε, ευρωπαϊκούς, όχι όλους, αλλά σε κάποιους, είδαν ότι προσπαθούσαν να υλοποιήσουν τοπικούς κανονισμούς κανόνες μάλλον και πρότυπα και έτσι ε, αρνούνταν να τους ε, δεχθούν. Ότι δεν συμμορφούνταν δηλαδή ε, με την οδηγία για το καθαρό νερό. Το αναφέραμε και τώρα στην Προεδρία σήμερα και στην προηγούμενη. Και θα θέλαμε να δούμε αν μπορεί να υπάρξει κάποια διευκρίνηση γιατί σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ανεχτούμε ε, την εφαρμογή κάποιων τοπικών κανόνων που δημιουργούν απλώς ε, σύγκρουση μεταξύ δύο διαφορετικών ε, κανονισμών ή οδηγιών. Δεύτερη παρατήρηση για τη ρήπανση. Το κύριο που ακούμε είναι εντάξει αν έχουμε μια πετρελοκυλίδα, κάποια μεγάλη καταστροφή. Μόνο τότε τα ακούμε αυτά. Βέβαια όμως ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που άπτονται τη ρήπανση σήμερα είναι τα πλαστικά και τα απόβλητα. Και δεν μιλάω μόνο για τα ε, σκάφη, γιατί εκεί έχουμε ξεκάθαρους κανόνες. Αλλά αν δείτε τα κράτη-μέλη ε, που πρόκειται ξεκάθαρα για ε, κράτη-μέλη που έχουν λιμάνια, και τον όγκο των απορριμμάτων που βγαίνουν μετά στη θάλασσα. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Μιλούμε για όλα αυτά τα γαλάζια και καθαρά ύδατα, όμω είναι μια τεράστια πρόκληση σε όλο τον κόσμο. Και με τη δική σα ε, ιδιότητα, που έχετε και μια συνολική εικόνα, διερωτώ με κατά πόσο ο δικός σας οργανισμός έχει ε, ιδέες και προτάσεις για το πώς μπορούμε να ε, καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο μαζί και παράλληλα με τα όσα κάνετε για τυχόν πετρελοκυλίδες κτλ. Αυτά από πλευρά μου. σα ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που σα ξαναβλέπω. Merci. Ευχαριστώ. Η κυρία Μοντέρο έχει το λόγο. Που είδαμε και στη φωτογραφία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Μιλή. Λυπάμαι που έχασα την εισήγησή σας αλλά ήμουν στην Επιτροπή Αλίας που λάμπανε χώρα την ίδια στιγμή. Θέλουμε όμως ε, και εμείς ε, να αυξήσουμε αυτές τις ε, επιτόπιες επαφές με τους επιτόπιους ελέγχους, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για ό,τι συμβαίνει. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. για ένα κοινό για την Ευρώπη ζήτημα, το προσφυγικό. Θα ήθελα όμως να σταθώ σε δύο σημεία και δεν θα ήθελα τα σχόλιά σας. Πρώτον, για το θαλάσσιο πακέτο που εξετάσαμε σήμερα το πρωί για την ασφάλεια των επιβατών που μας παρουσίασε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό άπτεται και του ρόλου της ΕΜΣΑ στις επιθεωρήσεις ε, των σκαφών. Εσείς λοιπόν πώς εκτιμάτε αυτή την προσέγγιση ε, βάση κινδύνου στις επιθεωρήσεις, όπως ε, συμβαίνει με την ε, οδηγία κράτους λεμένα. Μπορείτε να το σχολιάσετε το παρακαλώ. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για το θείο, πώς μπορεί να γίνει η πραγματικότητα. πώς μπορούμε να επενδύσουμε στο υγροποιημένο φυσικό αέριο ως ε, λιγότερο ρηπογόνο καύσιμο, το οποίο θα μας ε, επιτρέψει να ε, ρίξουμε, να μειώσουμε τις εκπομπές θείου. Και πώς θεωρείτε ότι προχωράμε σε αυτό το τομέα με βάση τις επιθεωρήσεις σας. Ο κύριος Ρίκε. Ευχαριστώ. Κύριε Διευθυντά, έχετε δει ότι η Επιτροπή μας εξακολουθεί να στηρίζει ευρέως τον οργανισμό σας και μετά την διεύρυνση των καθηκόντων σας. Υπάρχει ένας προβληματισμός, μια ανησυχία σε ό,τι αφορά τους υλικού και ανθρώπινους πόρου. Όμως ε, και ένα άλλο σημείο προβληματισμού το οποίο θα ήθελα να θίξω. Με τα νέα καθήκοντα σε ό,τι αφορά ε, την φύλαξη των συνόρων, εσείς θεωρείτε ότι έχετε ε, τα απαραίτητα κανονιστικά και ρυθμιστικά μέσα για να φέρετε εις πέρα στο έργο σας, εφόσον ο Frontex που επωφελείται κατά κάποιον τρόπο των πόρων σας δεν έχει ε, κανονιστική ε, πρόσβαση στην φύλαξη των συνόρων. Αυτό επηρεάζει τον τρόπο λειτουργία σας. Χρειάζεστε ρυθμιστική βελτίωση ή διεύρυνση της ε, νομοθετικής εξουσίας του οργανισμού σας. Θεωρείτε ότι το υφιστάμενο, δηλαδή κανονιστικό πλαίσιο, είναι επαρκές. Ευχαριστούμε κύριε Ρίκε. Ένα μικρό ερώτημα. Τον Φεβρουάριο του 2017 θα γίνει μια πρόσκληση υποβολή ενδιαφέροντος για 10 εκατομμύρια ευρώ για την εποπτεία των θαλάσσιων συνόρων μέσω drones, μέσω ε, αυτών των ε, μη επανδρομένων αεροσκαφών. Ε, τι είδους ρήπανση θα είναι αυτή που θα σας απασχολήσει. Αυτό είναι το αντίστοιχο ερώτημα αυτό της κυρίας Φώστερ. Ποιο είδος μόλυνσης θα ε, εξετάζεται πιο συγκεκριμένα. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά ε, τους drones και πάλι, ε, ποιο θα είναι, ποια θα είναι η τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου για να διευκολύνουμε ε, την εποπτεία. Πολλές οι ερωτήσεις, τώρα ο λόγος σε εσάς. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αξιότιμες και αξιότιμοι ευρωβουλευτές για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις συνοψίσω, διότι υπήρχαν και ορισμένε που επικαλύπτονταν. Πρώτα, για τον ρόλο του οργανισμού ΕΜΣΑ και τη νομική βάση για τα όσα πράττουμε. Έχουμε πολύ σαφή εντολή του ΕΜΣΑ που βασίζεται στον ε, θεμελιώδη κανονισμό και στις αναθεωρήσεις του. Αυτό μα λέει τι είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε. Πρόκειται για τι λεγόμενε βασικέ λειτουργίε του οργανισμού, core tasks στα αγγλικά, οι οποίε κυρίω έχουν σχέση με την ασφάλεια τη ναυσιπλοείας, προστασία του περιβάλλοντο και ζήτημα, ζητήματα μάλλον παρακολούθησης, Έρχομαι τώρα στη συνεργασία με τον οργανισμό Frontex και τον ΕΦΚΑ. Έχουμε διεξαγάγει συνεργασία μαζί τους για πολλά χρόνια. Και στο επίπεδο της διμερούς συμφωνίας και με τους δύο τους οργανισμούς έχουμε εδώ και καιρό, διότι η ΕΜΣΑ έχει την ικανότητα να παρακολουθεί θαλάσσιες περιοχές που δεν έχουν οι δύο αυτοί οι άλλοι οργανισμοί. Και δεν είναι ορθό να επικαλύπτονται τα συστήματα. Δεν είναι σκόπιμο. Γι' αυτό παρέχουμε σε ΕΦΚΑ και Frontex όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που, που έχουν ανάγκη. Και αυτοί όταν σε ορισμένα project ΕΦΚΑ και Frontex ή και πιο μακροπρόθεσμα για τον Frontex. Έχουμε για την ώρα τέσσερις υπαλλήλου του Frontex που έχουν γραφεία στον ΕΜΣΑ και αποκτούν εικόνα για τα συστήματα του ΕΜΣΑ. Διότι πρόκειται για ειδικέ πληροφορίε που συλλέγονται από τον ΕΜΣΑ. Όμως δεν τους αρκούν έτσι λοιπόν αναλύουν περαιτέρω τις πληροφορίες αυτές και μετά τις εντάσσουν στο ε, οικειοσύστημα. Άρα μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα που κάνουμε με, περισσότερο, με περισσότερη αποτελεσματικότητα χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες και των τριών οργανισμών. Για την υπόθεση της ακτοφυλακής είπα ήδη ότι ο ΕΜΣΑ οι περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες ακτοφυλακής είναι, συναποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων μας μπορούμε να πούμε ότι μας επιβάλλει κάπως περισσότερη εργασία, επειδή όμως ήδη είναι τμήμα των θεμελιωδών δραστηριοτήτων μας, δηλαδή και ε, η επιβάρυνση, ο έξτρα φόρτος εργασίας δεν είναι τρομερός. Είναι όμως σημαντικός εμπλουτισμός και όπως είδατε από το διάγραμμα, πρόκειται να απασχολήσουμε 17 πρόσωπα παραπάνω που <clears throat> θα, που θα ε, προσληφθούν ειδικά για αυτήν την υπηρεσία Coast Guard Function. Και μεταξύ άλλων θα αναπτύξουν και άλλο την συλλογή πληροφοριών μέσα στα συστήματα παρακολούθησης. Ρωτήσατε επίσης αν υπάρχουν εμπόδια, κολλήματα νομικά ή αν θα μπορούσε κάτι να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ο πολιτικός κόσμος. Υπάρχουν. Εμείς, μπορώ να πω, συζητούμε με αυτές τις ε, συζητούμε και με αυτά τα συστήματα παρακολούθησης και με την ΕΑΣΑ για να δούμε πώς μπορούμε να στείλουμε τα μη επιδρομένα αυτά αεροσκάφη σε ορισμένες περιοχές. Όχι όμως πάνω από την ξηρά και σε κατοικούμενες περιοχές. Μόνο πάνω από θαλάσσιες περιοχές. Γιατί αυτό είναι και το τμήμα, το τμήμα, το, ο τομέας των αρμοδιοτήτων μας. Και το όριο είναι βεβαίως η ακτογραμμή για μας. Δεν έχουμε όμως κανονισμό και αυτό αποτελεί ένα εμπόδιο και μια σημαντική πρόκληση για μας. Όπως είπα πριν, του χρόνου θα πρέπει να αρχίσουμε κανονικά να προσφέρουμε υπηρεσίες σε οργανισμούς και χώρες μέλη σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες μη επανδρομένων αεροσκαφών. Αυτό είναι πρόκληση για μας, γιατί θα πρέπει να πάμε σε κάθε χώρα μέλος να διαπραγματευτούμε με τις αρμόδιες αρχές πολιτικής αεροπορίας την άδεια να πετάξουν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μας. Τώρα, νέα υπηρεσία την οποία προωθούμε. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα drones με διαφόρους τρόπους. Θα κάνουμε την υπηρεσία αυτή μη επιδομένων αεροσκαφέων όσο γίνεται πιο αποτελεσματική. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε ορισμένες περιοχές με δορυφόρους, με AIS, αλλά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη θα παίζουν συμπληρωματικό χαρακτήρα, άρα θα προσθέτουν αξία στις υφιστάμενες, συστήματα συλλογής προφοριών μας θα εμπλουτίζουν τις πληροφορίες που συλλέγουμε ήδη. Άρα πρέπει να αναπτύξουμε και αεροσκάφη με πολλαπλούς αισθητήρε. Αυτό αποτελεί πρόκληση και για τους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συμβαλόμεθα και για τον ΕΜΣΑ. Και χρειαζόμαστε και την ενίσχυσή σας. Ο Κιθ Τέιλορ με ρώτησε για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου και τον ρόλο της ΕΜΣΑ ή του ΕΜΣΑ. Η λειτουργία ακτοφυλακής και άλλες δράσεις ρωτάτε εάν είναι μεγαλύτερη πρόκληση όλα αυτά για τους πόρους οικονομικούς και ανθρώπινους του ΕΜΣΑ. Είπα ότι περιορίζουμε το προσωπικό μας μετά από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περικοπές της τάξης 10%. Και τώρα, επειδή προστίθεται η ακτοφυλακή, προσλαμβάνουμε 17 πρόσωπα, άρα δηλαδή βρισκόμαστε λίγο πολύ στα ίδια, όπως, με, όπως το 2012. Τώρα, μετακινούμε το προσωπικό σε διάφορες άλλες υπηρεσίες για να μπορέσουμε να δώσουμε ανθρώπους που χρειαζόμαστε για αυτές τις ε, ειδικέ, τις εξειδικευμένες υπηρεσίες, δηλαδή εμπειρογνώμονες. Η εντολή που διαθέτουμε σήμερα δεν μπορεί να διευρυνθεί άλλο χωρίς να προβλεφθούν έξτρα πόροι, ανθρώπινοι και οικονομικοί, δημοσιονομικοί. Έχουμε φτάσει στα όρια. Μπορούμε να αποδώσουμε το έργο που ζητούν οι χώρες μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα stakeholder, δηλαδή τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας. Αλλά αρχίζουμε σιγά σιγά τώρα να βλέπουμε και τα όρια μας και κάποια εμπόδια. Και βλέπουμε ακόμη ότι από διάφορες πλευρές υπάρχει θέληση να ανατεθούν και άλλα καθήκοντα στον ΕΜΣΑ. Είδαμε τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος αλλά και τη Γενική Διεύθυνση Κλίματος που θα ήθελαν να διαθέτουν υπηρεσίες του ΕΜΣΑ για δική τους χρήση. Γιατί μπορούμε να τους προσφέρουμε και να εμπλουτίσουμε τις πληροφορίες που διαθέτουν μέσω των υπηρεσιών μας. Το θέμα του προσφυγικού, που είναι μέγα θέμα και όπου ο ΕΜΣΑ έχει ένα ξεκάθαρο ρόλο. Προσφέρουμε υποστηρικτικές πληροφορίες στον Frontex δεν αναλαμβάνουμε έξτρα ευθύνες στον τομέα αυτό. Διαθέτουμε όμως πληροφορίες, εμπλουτίζουμε πληροφορίες το έργο του Frontex και με τις δυνατότητες που έχουμε, όπως για παράδειγμα μία επαναδομένα αεροσκάφη αλλά και άλλα, προσφέρουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται το Frontex. Μπορούμε και δορυφορικά να βρούμε και μικρά σκάφη και βαρκούλες είναι καλή ικανότητα που προσφέρουν οι δορυφόροι. Ανακάλυψαν για παράδειγμα οι δορυφόροι μας ε, φουσκωτές βάρκες που, ε, μέσα στις οποίες βρίσκονταν 30 άτομα. Η ΕΜΣΑ, η δεν αναλαμβάνει άλλες δράσεις, προσφέρει μόνο τα δεδομένα αυτά στις αρμόδιες αρχές. Μετά συζητήσατε και το θέμα των εκπομπών θείου. Επ' αυτού μπορώ να πω ότι ο ΕΜΣΑ ήδη από τον αρχών του 2015 όταν άρχισε να ισχύει η οδηγία περιθείου συνεργαζόμαστε με τις χώρες μέλη και συλλέγουμε πληροφορίες για τις επιθεωρήσεις θείου σε περιοχές ΣΕΚΑ. Την πρώτη φορά 7.000 επιθεωρήσεις με συλλογή δεδομένων ο κλάδος εξεπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την οδηγία για το θείο. Αφενός αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι μειώθηκε πολύ η τιμή του καυσίμου. Μπόρεσαν λοιπόν να χρησιμοποιήσουν θαλάσσιο δίζελ με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα θείου. Ορισμένοι δε εφοπλιστές αποφάσισαν να εγκαταστήσουν και συστήματα καθαρισμού των καυσαερίων. Κάτι το οποίο βέβαια προκάλεσε και προβλήματα, όπως είπε και η κυρία Φώστερ με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Καθαρών Νερών, διότι αυτό προκάλεσε προβλήματα αφού τα νερά αυτά δεν μπορούσαν να διοχετηθούν στο θαλάσσιο νερό, στη θάλασσα δηλαδή, και έπρεπε να ε, ε, αποθηκευτούν σε λιμάνια, τα οποία δεν είχαν πάντα την κατάλληλη υποδομή. Πλαστικά και άλλα απορρίμματα. Για την ώρα δεν για τις αρμοδιότητές μας. Είναι και πολιτικά ευαίσθητο το θέμα, άρα θα χρειαστούμε πρώτα πολιτική απόφαση. Και πρέπει να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. LNC. Και οι σχετικές υποδομές που για το LNG, δηλαδή το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Ε, εκεί βεβαίως ε, χρειάζονται εγκαταστάσεις. Ορισμένα πλοία έχουν να ναυπηγηθεί που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και θαλάσσιο τίζελ αλλά και εναλλακτικά υγροποιημένο φυσικό αέριο αλλά χρειάζεται χρόνος μέχρι να υπάρχουν εγκαταστάσεις, να γνωρίζουν, ότι, να γνωρίζουν και οι ενδιαφερόμενοι ότι υπάρχουν σχετικές υποδομές και στα λιμάνια και χρειάζεται και πολύ περισσότερος χρόνος και στο παγκόσμιο επίπεδο. Σκεφτείτε, θα χρειαστεί να διέρχονται και τον Ατλαντικό. Οπότε η bunkering facilities δεν είναι επαρκής για την ώρα. Για θέματα ασφάλειας τώρα, που είναι βέβαια κάτι το οποίο προωθείται πολιτικά πολύ. Η, ο ΕΜΣΑ κάνει τις επιθεωρήσεις, είναι θέμα αρμοδιότητός μας, συνεργαζόμαστε και με τον ε, Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοείας. Θα δούμε τι θα προκύψει από τον επόμενο MSC για την ασφάλεια των επιβατών, επιβατικών, επιβατικών πλοίων. Αυτά λίγο πολύ με ρωτήσατε. Εάν παρέλειψα κάτι, παρακαλώ υπενθυμίστε το μου. Ίσως μπορώ να τονίσω για μια φορά ακόμη τον κανονισμό για τα μη επιδομένα αεροσκάφη. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μπορεί ο ΕΜΣΑ να χρησιμοποιήσει την σύγχρονη τεχνολογία και στο μέλλον και χρειαζόμαστε εναρμονισμένο κανονισμό που να προέλθει από το ευρωπαϊκό επίπεδο για να διευκολύνει το έργο μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, λέει ο Πρόεδρος, για να σας διευκολύνουμε όσο μπορούμε περισσότερο από την πλευρά της δικής μας Επιτροπής. Σας ευχαριστώ λοιπόν που προσήλθατε εδώ. Μας τα είπατε με αρκετή ακρίβεια, μας δώσατε πολλά στοιχεία. Πάντοτε θα μπορείτε να βασίζεστε στην υποστήριξή μας μέσα στην βούληση να ενισχύσουμε το ρόλο του ΕΜΣΑ που βεβαίω αντιμετωπίζει σημαντικέ προκλήσει. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε λοιπόν με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, την έκθεση της κυρίας Κιουλόνεν. Υποχρεωτικές μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 2021 με 2030. Κυρία Κιουλόνεν, έχετε το λόγο για την παρουσίαση της εκθέσεώς σας, της πρότασης γνωμοδότησής σας μάλλον. Και μετά θα δώσω το λόγο στους Σκιώδης. Και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχετε το λόγο κυρία Κιουλόνεν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους για το ενδιαφέρον τους Ήταν ιδιαίτερα θετικό το, οποίο, το ότι μπορέσαμε να πάρουμε την Επιτροπή αυτή και εξ ονόματος Επιτροπής Περιβάλλοντος ήδη από το 1990 έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις για τη μείωση των εκπομπών καυσαερίων ε, τις μεταφορές. Το θέμα αυτό έχει τεθεί επανειλημμένα υποσυζήτηση, αλλά δυστυχώς ε, οι εκπομπές αυξάνονται. Το 2014 ήταν 20% υψηλότερες από ό,τι το 1990. Στόχος λοιπόν αυτής της νομοθετικής πρότασης είναι να καλύψει το σύνολο του τομέα εκτός από τις θαλάσσιες μεταφορές και τις αερομεταφορές. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση κανονισμού, τα κράτη-μέλη καλούνται να μειώσουν τις εκπομπές από το, από το 2020 μέχρι το 2030, 2021 ε, μάλλον 2030, επί τη βάση εθνικών ποσοστώσεων και γραμμικών μειώσεων για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο λοιπόν εγώ προσπάθησα να κάνω ε, για τους στόχους μείωσης οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2030 η βασική ιδέα είναι η συμφωνία αυτή κατανομής των βαρών να συνδεθεί και με τη Συμφωνία των Παρισίων και με τις ευρύτερες ανηλυμένες υποχρεώσεις για μείωση εκπομπών. Η περίοδος 21-30 σημείο εκκίνησης είναι μάλλον το 2020 και θα χρησιμοποιηθεί σαν βάση το σύνολο των στοιχείων που θα παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 16-20. Θα πρέπει να υπάρξουν ε, αντίστοιχες, ε, αντίστοιχα κίνητρα για όλες τις χώρες για να μειώσουν τις εκπομπές και γι' αυτό λοιπόν προτείνω τα, 2000, τα επίπεδα του 2020 να αναθεωρηθούν προς τα κάτω. θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη μας ε, το μέσο όρο 16-20 ή τις τελευταίες επιδόσεις το 2020. Μιλάμε για 93 μεγατόνους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεριλάβει στην πρότασή της συγκεκριμένα στοιχεία για την αποτελεσματική χρήση των μέσων κάποια στοιχεία ευελιξίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια κατάσταση στα πλαίσια της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να τηρήσει τις υποχρεώσεις ε, και τους στόχους των Παρισίων. Το επίπεδο παραδοχής ε, στα κράτη-μέλη εξαρτάται κυρίως από την ίδια, αν θέλετε, αυτή την ευελιξία εκεί όπου δικαιολογείται η ευελιξία θα μπορούσε να υπάρξει ένας μηχανισμός άπαξ χρησιμοποιούμενος päästövähennyspolku pysyisi jäsenmaissa hallittuna.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 θα πρέπει να γίνεται ετήσια αξιολόγηση για το πώς πετυχαίνουμε τους στόχους στην ουσία γιατί νομίζω ότι η πενταετής αναθεώρηση δεν είναι επαρκής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει σαφή μέσα και να είναι σε θέση να επιβάλλει κυρώσεις εις βάρος των κρατών μελών που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Τώρα, ειδικά για τις μεταφορές, θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζω την πρόταση στα πλαίσια της οποίας οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη. Έχω την εντύπωση όμως ότι είναι, ότι θα ήταν μάλλον προβληματικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει τον συντονιστικό ρόλο ο οποίος θα της επέτρεπε να εφαρμόσει τις βέλτιστες πρακτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα ειδικά χρηματοδοτικά της μέσα θα μπορούσε να είναι σε θέση να κατανείμει μια σημαντική σειρά χρηματοδοτήσεων και οι χρηματοδοτήσεις αυτές θα πρέπει να στοχευθούν και στον τομέα των μεταφορών προωθώντας μια μεταβατική περίοδο σε συστήματα μεταφορές χαμηλών εκπομπών ή και ελευθέρων από εκπομπές μεταφορικών συστημάτων. suunnittelusta, Νομίζω λοιπόν ότι εδώ θα μπορέσουμε να προωθήσουμε δυνατότητες όπως ε, το βάδισμα, η ποδηλασία, να χρησιμοποιήσουμε επίσης νέα συστήματα χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων, όπως επίσης και τιμολογιακά μέσα για να ευνοήσουμε τη χρήση συγκεκριμένων μέσων. Αυτό θα επιτρέψει την δημιουργία νέων μέσων κινητικότητας, έτσι ώστε οι πολίτες να εγκαταλείψουν τα μεμονωμένα οχήματα και αυτό να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για το μέλλον. Είναι επιθυμητό οι νέες αυτές υπηρεσίες να καταστούν λειτουργικές ε, για την κάλυψη αναγκών των αστικών και περιαστικών περιοχών, να διευκολύνουν τις μετακινήσεις και να καταστήσουν το κόστος των μετακινήσεων διαφανές και προβλέψιμο. Οι αυτοματισμοί στον τομέα των μεταφορών προχωρούν ταχύτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί στο παρελθόν, ως εκ τούτου αυτά τα θετικά σημεία δίνουν την δυνατότητα στους νομοθέτες στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθήσουν από κοντά το πόσο επηρεάζουν ε, το επίπεδο των εκπομπών. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν θα είναι πιο ευνοϊκά για το κλίμα και το περιβάλλον ιδιαίτερα σε επίπεδο τοπικό. Οι μετακινήσεις των Ευρωπαίων πολιτών είναι από τις πιο σημαντικές παρεχόμενες υπηρεσίες σε καθημερινή βάση. Επακριβής και ε, ελεγχομένου κόστους ε, επιμελητιακές υπηρεσίες είναι επίσης χρήσιμες και για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Στα πλαίσια λοιπόν του προγράμματος κατανομής του βάρους έχουν καθοριστεί φιλόδοξοι στόχοι και εγώ εδώ θα ήθελα να μου επιτρέψετε να εκφράσω και την ανησυχία μου, διότι το κόστος της μεταφορικής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων στην Ευρώπη γενικά δεν είναι κάτι το προβλέψιμο. Ένας υπολογισμός αξιόπιστος ωφέλους μπορεί να γίνει μόνο μετά την κατανομή των υποχρεώσεων μείωσης εκπομπών. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δώσει τα απαιτούμενα μέσα στα κράτη-μέλη. Ελπίζω η συζήτηση να είναι ενδιαφέρουσα και να συνεχίσω τη συνεργασία με τους Κιώδης. Ευχαριστούμε κυρία εισηγητρία. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στους Κιώδης συζητητές. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για τις προτάσεις της. Έχει δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για τη συνεργασία μας και την ευχαριστώ. Χαιρετίζω και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έγγραφο και χρειάζεται συλλογική προσπάθεια από όλα τα κρατημέλη για να διασφαλίσουμε την επιτυχή αυτή μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλή κατανάλωση άνθρακα. Και με την πρόταση προβλέπονται ξεκάθαροι κανόνε ε, για να διευκολυνθεί αυτή η μετάβαση. Βεβαίω θέλουμε να δώσουμε και νέε ευκαιρίε για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη, ενώ θα μετριάσουμε ε, την τη ζημία από ε, την κλιματική αλλαγή, έχουμε και τα ελάχιστα ε, όρια που πρέπει ε, να επιτευθούν μέχρι το 2030 και τη δέσμευση των κρατών μελών να περιορίσουν τις εκπομπές του, των αερίων του θερμοκηπίου. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις επιμέρους και διαφορετικές δυνατότητες των κρατών μελών και έτσι να θέσουμε διαφορετικούς στόχους ανάλογα με το κατακεφαλήν ΑΕΠ. Νομίζω ότι έτσι διασφαλίζεται η δίκαιη αντιμετώπιση, γιατί οι χώρες με υψηλότερα εισοδήματα μπορούν πιο εύκολα ε, να υλοποιήσουν αυτές τις εφαρμογές. Μπορούν από κοινού κάποια κράτη-μέλη να ε, μειώσουν τις εκπομπές τους με βάση τις ε, επιχειρηματικές δραστηριότητε και για την ευελιξία. Αρχικά έχουμε ευελιξία σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις πιστώσεις, ε, από τον τομέα χρήσης γης και από τις πιστώσεις για τις εκπομπές. Θα υπάρξει υποχρέωση ε, συμμόρφωσης και υποβολής εκθέσεων και τα έχει αναφέρει αυτά και η συγκίτρια. Και ξέρω ότι θα τα συζητήσουμε αυτά όταν περάσουμε ε, στα επιμέρους της υποβολής εκθέσεων. Πάντα θέλουμε να βρούμε τρόπους αύξησης της ενεργικής απόδοσης το 75% των εκπομπών ε, των αερίων του στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκύπτει ακριβώ από αυτό. Ε, Στι μεταφορέ ε, πολλά μένουν ακόμα να γίνουν, βέβαια. Θέλουμε ευφυείς, βιώσιμε τεχνολογίες που θα μας ε, βοηθήσουν ε, να συνεχίσουμε αυτή την οδό. Θέλουμε να παραμείνουμε ε, ηγέτιδα δύναμη στα, στις ανταγωνιστικές αγορές και στις υπηρεσίες, όμως πρέπει να διατηρήσουμε κάποια ισορροπία, γιατί και τα τιμωρητικά μέτρα δεν οδηγούν σε συνεργασία ε, και την επίτευξη συλλογικών στόχων. Δεν πρέπει λοιπόν να λειτουργούμε τιμωρητικά σε τεφορά του κοινού ε, στόχου. Δεν πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα επιβάλλει ε, διορθωτικά μέτρα χωρί καμία εγγύηση θετικού αποτελέσματο. Πρέπει να υπάρχει αυτή η ισορροπία μέσα στο κείμενο. Βέβαια, η αρχή της ευελιξίας παραμένει η βασική αρχή της πρότασης της Επιτροπής και προκύπτει και από το κείμενο των Παρισίων. Χαιρετίζουμε λοιπόν τις προτάσεις και προσβλέπω στη συνεργασία μας με την εισηγήτρια προκειμένου να υποβάλουμε μια συλλογική πρόταση στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γοηβό Ντελόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την εισηγήτρια κυρία Κιλόνανεν για την ε, πρώτη αυτή παρουσίαση. Ως ασκιώδης ε, από πλευράς σοσιαλιστών δημοκρατών θα ήθελα πάνω απ' όλα να επισημάνω πόσο σημαντικό είναι το κείμενο που εξετάζουμε σήμερα. Πρόκειται για την ε, μετάφραση ε, και μεταφορά του κειμένου των Παρισίων σε ευρωπαϊκό δίκαιο. Θα είναι το θεμελιώδες πλαίσιο σε ό,τι αφορά του ε, στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή για τα επόμενα 30 χρόνια. Από αυτή την άποψη θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο τη, γιατί ενισχύει την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν είχε επαρκή επίπεδα φιλοδοξία. Πρώτον, η συμπερίληψη κλιματικών στόχων για το 2050 είναι πολύ σημαντική για να εγγράψουμε, για να εξετάσουμε μάλλον την ευρωπαϊκή δράση πιο μακροπρόθεσμα όπω προκύπτει και από το Παρίσι. Είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε την ε, διαχείριση στόχων προτείνοντα ε, έναν πιο συστηματικό έλεγχο συμμόρφωση και συμπεριλαμβάνοντα μια πραγματική ρήτρα αναθεώρηση. Για να συμπληρώσω αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης θα έχω αρκετές προτάσεις για να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο το επίπεδο φιλοδοξιών του κειμένου. Για να μην υπάρχει δωρεάν κατανομή των πιστώσεων, καλό θα ήταν να ισχύσει το, ένα αντίστοιχο σύστημα με το ETS, δηλαδή ε, ε, ετησίως να γίνεται... Ε, να ευνοηθεί η αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Μετά για τη ρήτρα αναθεώρηση, καλό θα ήταν να ενισχύσουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντο σε ό,τι αφορά του κλιματικού στόχου. Ε, πρέπει να περιορίσουμε ε, τη δυνατότητα ευελιξία που παρέχεται σε κάποια κρατη κράτη-μέλη. Θα ήταν απαραίτητο, κατά τη γνώμη μου, να αναθεωρήσουμε το σημείο εκκίνηση σε ό,τι αφορά την πορεία μείωση ε, των εκπομπών, ούτω ώστε η κατανομή των ποσοστώσεων να μην υπερβαίνει σε μεγάλο βαθμό τι πραγματικέ εκπομπέ των κρατών μελών κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται ίσονο σημασία, νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε και τον τίτλο. Να είναι πιο σαφή ε, και να, ε, δίνει, να προκαλεί το ενδιαφέρον των πολιτών για να καταστεί πιο ευανάγνωστο. Ευχαριστούμε ο κύριος ε, Τέλτσικα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αρχίσω λέγοντας ότι και νομίζω συμφωνούμε. Σημαντικό, σημαντικό θέμα. Χρειαζόμαστε ισορροπία και χρειάζεται και ένα χαρακτήρα που να μην αποκλεί κανένα. Συμφωνώ με τα όσα είπε η συγκητρία που μου φαίνονται ισορροπημένα. Είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξω και σε άλλα ε, σχόλια, αλλά βέβαια πρώτα θέλω να διαβάσω το σχέδιο. Ήδη τώρα επισημαίνω την τροπολογία 11 για το άθο 1, όπου η συγγήτρια μιλεί για την προσπάθεια επίτευξης των στόχων, για τους οποίους οι χωρισμένοι θα πρέπει να συνεχίσουν να μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηρυπίου κλπ. Και βάζει τους στόχους για 2030, 40, 50. Κατανοώ την φιλοδοξία των στόχων και ευχαρίστως να συμφωνήσω. Διερωτώ με όμως εάν αυτά ακριβώς θα μπουν στο σχέδιο κανονισμού με την έννοια ότι τα νούμερα αυτά είναι σε πολύ μακρινές ημερομηνίε και μα ίσως μάλιστα να τα πάμε και καλύτερα, ίσως να αντιμετωπίσουμε άλλα προβλήματα. Γι' αυτό προσπαθώ να είμαι πάντοτε ακριβής σε θέματα ημερομηνιών και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να ρωτήσουμε πρώτα το τμήμα EPRS που κάνει έρευνες για λογαριασμό των βουλευτών. Δεν αμφισβητώ την ισχύ της προτάσεως, δεν αμφισβητώ την ορθότητα της προτάσεως, αλλά διαρωτώ με εάν είναι ίσως υπερβολικά φιλόδοξη. Νομίζω ότι χρειάζεται μια επανεξέταση πριν από το 2030. Και μπορούμε ίσως ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή να ζητήσουμε μια μελέτη αντικτύπου. Για την τροπολογία 9, για τους στόχους 2020 δηλαδή, που περιλαμβάνονται στην απόφαση, σε ό,τι αφορά την οδό που θα ακολουθηθεί. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να μπουν αυτά στη βάση των μέσων όρων 2016 έως 2018. Και διαβάζει το κείμενο. Much more significant efforts to reduce emissions uh, and have lower emissions in 2016 and 18. Νομίζω λοιπόν ότι το κείμενο αυτό δεν υποστηρίζει και την συνέχεια των προσπαθειών μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου. Όμως, ο λόγος που κρύβεται πίσω από την προσέγγιση αυτή είναι κατανοητός και ίσως μπορεί να υπάρξει ένα συμβιβασμός να μειωθούν δηλαδή οι, τα πιστοποιητικά στο επίπεδο των στόχων των χωρών μελών μέχρι το 2020. ανταμείβοντας έτσι τις αρχικές προσπάθειες που έγιναν για τη μείωση του πλεονάσματος AA. Έχω και την τροπολογία 10 για την παράγραφο 3 του άρθρου 5 για το 5% δεν μου προκαλεί κανένα μεγάλο πρόβλημα. Διαρωτώ με όμως, εάν δεν μπορούμε να δώσουμε κίνητα στι χώρε μέλη να κάνουν κάτι παραπάνω. Δεν είμαι και βέβαιος για το αν πράγματι θα έχουν αντίθετο αποτέλεσμα από το αναμενόμενο. Ή αν οι χώρες μέλη θα κάνουν μια έξτρα προσπάθεια. Και πόσο πιθανό είναι. 5% λοιπόν μέγιστο όριο μεταφοράς σε άλλη χώρα μέλος. Πάντως εγώ ευχαρίστω να το εξετάσω και να δούμε πώς μπορεί. Την τροπολογία 8 δεν καλύπτεται εδώ, τροπολογία 11 που είναι και η τελευταία μου παρατήρηση. Η πρόταση να διαγραφεί στο 2027 και το 2032 για τις εκπομπές αερίου θερμοκηπίου κλπ. Η συμμόρφωση μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη ή θα είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί με τα μέτρα ευελιξίας. Και για το ποσό 1,08 και αν θα μειωθούν υπερβολικά τα AA και θα είναι δύσκολο να επιτευχθούν. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι υλοποιήσιμο κάτι τέτοιο και αν χρειάζεται διόρθωση για το σχέδιο της Κομισιόν. Αλλά αξιολόγηση αναδιαιτία περίπου νομίζω μπορεί να ικανοποιήσει την εισηγητέα και να είναι ταυτόχρονα και υλοποιήσιμο. Και εσύ κυρία εισηγητέα και εσείς κυρία Πρόεδρε είχα και άλλες παρατηρήσεις αλλά για να μην χάνουμε περισσότερο χρόνο, θα υποβάλω συγκεκριμένες διατυπώσεις σε συνεργασία και με τους άλλους σκιοδησιητές. Βέβαια, θα επανεξετάσω τις επιπτώσεις των όσων προτείνει η εισηγήτρια, ώστε να έχουμε μια στέρεα βάση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Κιφ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ε, είναι κοντά μας ο Μπάς Χάουτ, γι' αυτό και επειδή δεν του μοιάζω τόσο πολύ, θα, δεν θα προσπαθήσω να τον παραστήσω, αλλά θα μεταφέρω μόνο τα σχόλιά του, αφού ευχαριστήσω πρώτα την εισηγήτρια, που η εισήγησή της περιέχει ορισμένα καλά στοιχεία βελτίωση της προτάσεως της Κομισιόν πρώτα, εξασφαλίζοντας ότι χώρες οι οποίες δεν πληρούν τους στόχους του 2020 δεν επιβραβεύονται κιόλας από πάνω. Τροπολογία 12 για παράδειγμα στην έκθεσή σας που λέει ότι η χώρα μέλος θα πληρώνει 100 ευρώ για κάθε τόνο ισοδύναμου ε, διοξιδίου του άνθρακος πάρα που θα, που θα ε, παραπάνω. Τώρα για τις χώρες εκείνες οι οποίες ε, τηρούν τις δεσμεύσεις, η πορεία των μειώσεων δεν δείχνει ποια θα είναι μέχρι το 2021. Εμείς θα καταθέσουμε και τροπολογίες για να διασφαλίσουμε ότι οι χώρες μέλη δεν θα οδηγηθούν σε έναν διωγγωμένο Προπολογισμό ε, από την αρχή ήδη του εγχειρήματο. Ούτε η κλείνει τα κενά του συστήματος εμπορίας ε, των ε, εκπομπών η πρόταση της συγκεκριάς. Θα πρέπει όλοι να παίξουν τον ρόλο τους για την μείωση των αερίων. Το να χρησιμοποιηθούν τώρα τα πλονάσματα των ETS από την ε, μη ε, διαρκή χρήση των γιών και να αφήνουμε απ' έξω τον ε, το των μεταφορών είναι επικίνδυνο για το κλίμα και δεν δίνει κίνητρα για καινοτομία. Και εκεί λοιπόν να καταθέσουμε τροπολογίες για να διασφαλίσουμε ώστε τα διάφορα νομοθετήματα να παραμείνουν ξεχωριστά. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της έκρησης αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει βέβαια να διασυνδεθούν να συνδυαστούν. Τέλος θα πω ότι μας αρέσει η μείωση των πλεονασματικών πιστοποιητικών γιατί αυτό θα βελτιώσει την προσπάθεια επίτευξης των στόχων του 2030. Γνωρίζουμε όλοι τώρα ότι ο στόχος είναι πολύ χαμηλός. Αλλά αν θέλουμε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας που απορρέαν από τη συνθήκη του Παρισιού, ωστόσο αποτελούν ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Η πρόταση την οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρνητική. Δημιουργεί διακανονιστικού τύπου επιβαρύνσεις για τα κράτη-μέλη και τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις τους. Η έκθεση όμως την οποία προτείνεται είναι ακόμα χειρότερη διότι ιδεολογικοποιεί βλάπτοντας τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των οικονομικών κυρώσεων. Εσείς λέτε στους φτωχούς Ευρωπαίους ότι το κράτος του θα πρέπει να πληρώνει όταν μολύνουν πολύ ενώ οι ίδιοι δεν θα έχουν να φάνε. Η εφαρμογή του συστήματος αυτού είναι αμφίβολη ήδη και θέλετε εσείς την ευελιξία να την καταργήσετε ουσιαστικά, κάτι το οποίο είναι το μόνο που βοηθάει. Εσείς θέλετε επίσης η πενταετής επανεξέταση να γίνεται ετήσια. Όταν αυξηθεί ο διπλασιαστή ο αριθμός των ανέργων, τότε πραγματικά το ποδήλατο και ε, φυσικά το να περπατούν με τα πόδια θα χαροποιήσουν τους οικολόγους αλλά θα είναι και η μόνη λύση για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ο βασικός οικονομικός ανταγωνιστής μας είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε και επέλεξαν ένα πρόεδρο ο οποίος όπως ακούσατε αρνείται να εφαρμόσει τη Συμφωνία των Παρισίων, θα συνεχίσει ε, την εξόριξη φυσικού αερίου και πετρελαίου από σχιστόλιθο και θα ελαφρύνει τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς αυξάνοντας την αγοραστική ικανότητα ε, των Αμερικανών, μειώνοντας τις τιμές του κασίμου. Συνεπώς λοιπόν εσείς επιβαρύνετε τους κατοίκους μας, ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε απαλλάσσονται από τέτοιου είδους λογικές. Οπότε η ευρωπαϊκή παραγωγικότητα θα καταστραφεί. Όπως είπε ο Μαρκ Ρούτε, στον Ταβό την προηγούμενη εβδομάδα. Ξεχάστε τις ρομαντικές σας ιδέες, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για τη διάλυση της Ευρώπης. Το παράδειγμα του Brexit δεν σας αρκεί. Συνεχίζετε να επιλέγετε την ιδεολογία εις βάρος της πραγματικότητας και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα σας πεποιηθούν σύντομα. Je donne la parole à Monsieur Kramer. Ευχαριστώ. Δυστυχώς ήρθα με κάποια καθυστέρηση και δεν πρόλαβα να ακούσω όλη την παρουσίαση της ηγετίας. Βεβαίως καλούμεθα να την συζητήσουμε και όπως άκουσα μόλι, εάν δεν το κάνουμε τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Όταν μιλούμε λοιπόν για ανεργία ή για ποιότητα ζωής, όλοι αν θέλουμε να καταναλώνουμε και να μην κάνουμε τίποτα για την ε, ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ε, δεν θα ζήσουμε και πολύ και μπορεί να μιλήσουν και τα παιδιά και τα εγγόνια μα. Και αυτή είναι η ευθύνη που έχουμε απέναντι στι επόμενε γενναίε. Το άσχημο είναι ότι στον τομέα των μεταφορών καλούμεθα να κάνουμε πολλά, πάρα πολλά πράγματα, γιατί επί χρόνια, να μην πω δεκαετίες, έχει αγνοηθεί ο τομέα των μεταφορών, σαν να μην έχει καμιά σχέση με την αλλαγή του κλίματο. Ενώ είναι ο μόνο τομέα που έχει δει να ανεβαίνουν οι εκπομπέ των αερίων θερμοκηπίου από το 90 και μετά. Ενώ σε όλους τους άλλους τομείς καταφέραμε να τα μειώσουμε. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Για πολλά χρόνια, για να μην πω για πολλές δεκαετίες, η αυτοκινητοβιομηχανία με πραγματικά εγκληματικό τρόπο εξαπατά τον κόσμο και επιβαρύνει το περιβάλλον. Και η πρώτη αντίδραση της Κομισιόν ποια ήταν, άλλαξε τα όρια. Άλλαξε τα όρια. Δεν ήρθε να τους πει όχι πρέπει να τα τηρείτε παρόλο τον εγκληματικό τρόπο με τον οποίο είχαν εξαπατήσει όλο τον κόσμο. Ούτε ε, συνελήφθη κανείς, ούτε κρατείται, ούτε εξετάζεται. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ρεαλιστικές δοκιμές οι οποίες θα ελέγχονται και θα επιβάλλονται από ανεξάρτητους οργανισμούς. Αυτά πρέπει να τα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω και εμεί πρέπει να παίξουμε το ρόλο μα ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι χωρισμένοι. Για το εμπόριο των εκπομπών. Όταν το είχαμε πρώτο τότε είχαμε πει «Α, να, αυτή είναι η λύση διότι δίνεται υλικό κίνητρο, δηλαδή στις επιχειρήσεις για να μειώνουν τις εκπομπές». Όμως επειδή δόθηκαν πάρα πολλά δικαιώματα εκπομπής δωρεάν και μειώθηκαν τελικώς οι τιμές και η Ευρώπη δεν καταφέρνει επιτέλους να επιβάλλει μια ρεαλιστική τιμή, τα πράγματα συνεχίζονται. Και τα πράγματα συνεχίζουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και είναι πάντοτε φθηνότερο να εκπέμπουν απλώ τα καυσαέρια αυτά στην ατμόσφαιρα αντί να προσπαθούν να τα φιλτράρουν. Πρέπει λοιπόν να διδαχθούμε κάτι. Οι δε στόχοι του 2020 ωραία ήταν, θαυμάσια ήταν, αλλά θυμούμε ότι και σε αυτά οι μεταφορέ δεν έπαιζαν ρόλο. Η Κομισιόν είχε εγκρίνει στόχου μέχρι το 2020 υπό την κατεύθυνση τη καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ πάλι εκτός μεταφορών. Εμείς εδώ στην Επιτροπή μας είχαμε πει ότι πρέπει να συμβάλλει και ο τομέας των μεταφορών. 20% μείωση στην βάση των τιμών του 1990. Όμως το Συμβούλιο αρνήθηκε να συνεργαστεί. Ούτε ήθελε να το αγγίξει. Και όσο περισσότερο περιμένουμε, τόσο πιο μακρινή θα είναι η στόχη. Πρέπει να αρχίσουμε λοιπόν πολύ νωρίτερα και να είμαστε πιο φιλόδοξοι, διότι, παράδειγμα, γνωρίζετε ποια είναι η κατάσταση στην Κίνα που δεν έχω πάει τα τελευταία χρόνια, αλλά δέστε τι γίνεται εκεί. Οι Κινέζοι τουλάχιστον όμως τώρα είπαν, έχει καλώς, θα κάνουμε τις μεγαλύτερες επενδύσεις ανά τον κόσμο σε ανανεώσιμες ενέργειες. Αν εμείς τα καταφέρναμε έστω και το μισό να κάνουμε από αυτό που κάνουν οι Κινέζοι στις ανανεώσιμες ενέργειες, θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε κατά πολύ την κατάσταση του κλίματος. Πρέπει λοιπόν να διδασκόμαστε από το καλύτερο παράδειγμα και όχι από το χειρότερο, διότι έχουμε επιτέλους, όπως είπε, ευθύνη απέναντι στις μελλοντικές γενιές. Ευχαριστώ τον κύριο Κράμερ. Θα δώσω το λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που προσκαλέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ορισμένα σχόλια. Uh, Τρία σχόλια. Πρώτον, για θέματα φιλοδοξιών, δεύτερον, για θέματα ισοτιμίας και τρίτον, για θέματα ανταγωνισμού. Στο πρώτο, αυτό το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από πλευράς της Επιτροπής είναι ότι οι στόχοι, έτσι όπως έχουν συσταθεί εδώ και μέσω των τροπολογιών, δεν έχουν αξιολογηθεί σε σχέση με τις επιπτώσεις τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το οποίο έχουμε στο νου μας είναι να κάνουμε μία αξιολόγηση συνεπειών και για τους μακροπρόθεσμους στόχους, πέραν του 2030 δηλαδή, τα επόμενα χρόνια. Συνεπώς λοιπόν η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν θα πάρουμε τις τελικές αποφάσεις για το 2030 τώρα, αλλά σε μια υστερότερη φάση για την δικαιοσύνη και ισοτιμία, για την τροπολογία 13, όπου προτείνεται μια διαγραφή. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό άρθρο της πρότασης. Είναι ένα άρθρο το οποίο μας διασφαλίζει να μην υπάρχουν αντιφάσεις ανάμεσα στα διαφορετικά άρθρα και ιδιαίτερα στις χώρες χαμηλών εισοδημάτων όπως την Ανατολική Ευρώπη μέχρι το 20 να αυξάνουν και από το 20 και μετά να κατεβαίνουν. Αν εμείς βάζαμε το σημείο εκκίνησης το 2018 τότε στην ουσία θα διαγράφαμε αυτό το οποίο έχουμε ήδη νομοθετήσει και θα ήταν άδικο για τις χώρες αυτές. Γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε αυτή την συγκεκριμένη ρύθμιση. Το τελευταίο σημείο αφορά το διοικητικό βάρος. Αυτό αφορά τις αναφορές και την συμμόρφωση. Ίσως εδώ η πρόταση να μην είναι ξεκάθαρη. Αυτό το οποίο είναι σαφές και θα συμφωνήσουμε με τον εισηγητή, την εισηγήτρια μάλλον, είναι ότι είναι απαραίτητη η ετήσια παρακολούθηση, ο ετήσιος έλεγχος. Το θέμα είναι πότε θα γίνει ο έλεγχος συμμόρφωσης. Αυτή είναι μια επιπλέον διαδικασία, είναι μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία και εμείς ε, εδώ θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τις πέντε ετήσιες επιθεωρήσεις. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι αν μια χώρα δεν πετύχει τους στόχους της ένα συγκεκριμένο χρόνο, ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τις επόμενες πενταετής προβλέψεις γιατί ο έλεγχος συμμόρφωσης θα γίνεται συνεχώς επί ετήσιας βάσεως. Και αυτό το οποίο ε, θέλουμε να κάνουμε, είναι αυτό που κάνουμε έτσι κι αλλιώς μέχρι τώρα, είναι να δημοσιεύουμε ε, μια ετήσια έκθεση για τα κράτη-μέλη τα οποία οδεύουν στην επίτευξη των στόχων τους με πλήρη διαφάνεια έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να δουν αν θα αποτύχουν στην προσπάθειά τους ή αν πράγματι ε, θα τα καταφέρουν. Επίσης σε σχέση με τη χρήση γης και τη δασική παραγωγή και εδώ ο κύκλος αναφοράς είναι πενταετής κύκλος, οπότε κάθε πέντε χρόνια θα γνωρίζουμε πόσους πόντους θα παίρνει κανείς από τον συγκεκριμένο τομέα. Αυτό είναι δύσκολο να καταφέρει κανείς να το ελέγξει με τις ετήσιες μορφές επιθεώρησης που προτείνονται εδώ. Και πολλές από τις χώρες δεν θα γνωρίζουν τι credits θα έχουν, τι πόντους θα έχουν στη διάθεσή τους, αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη χρήση γης. Κάτι το οποίο θα καταστεί επίσης και ιδιαίτερα κοστοφόρο για τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε να το σκεφτείτε ξανά. Είναι μια καλή πρόταση που περιορίζει το διοικητικό βάρος για τα κράτη-μέλη. Μια τελευταία παρατήρηση. Η πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη για την ανάλυση κόστους-οφέλους, αυτό γίνεται εδώ και δύο-τρία χρόνια. Υπάρχουν συστηματικές ανταλλαγές απόψεων, στοιχείων και στα πλαίσια του χειμερινού πακέτου τα κράτη-μέλη καλούνται να προετοιμάσουν ε, προγράμματα δράσης για την ενέργεια. Συνεπώς δεν είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί εκ νέου και σε αυτήν την ομοθετική πρόταση. Σας ευχαριστώ και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας τις επόμενες εβδομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ. Άκουσα μία φράση η οποία έλεγε ότι η οικολογία είναι ιδεολογία. Η οικολογία δεν είναι ιδεολογία. Η οικολογία είναι μία πραγματικότητα και εδώ στις Βρυξέλλες ζούμε κάτω από κορυφές μόλυνσης και τα πρώτα θύματα των κλιματολογικών αλλαγών είναι οι πιο φτωχοί από τους συμπολίτες μας. Στόχος μας λοιπόν είναι όλοι να μπορέσουν να, προάγουν την ευημερία τους και την ποιότητα της ζωής τους και αυτό το οποίο ίσως έχει ξεχαστεί στον τομέα του COP21 είναι οι μεταφορές. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας κάνει μια πρόταση πάνω στην οποία θα γίνει μια έκθεση γιατί για πάρα πολλά χρόνια εμείς ήμασταν πρωτοπόροι στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης και θα πρέπει να ξαναγίνουμε το ταχύτερο δυνατόν. Μετά από αυτά τα λίγα λόγια θα δώσω το λόγο πάλι στον εισηγητή μας, στην εισηγήτρια μάλλον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς δεν ε, έχουμε εδώ σαν βασικό στόχο το απλά να σώσουμε μάλλον το πλανήτη ε, για τις επόμενες γενιές. Είμαι βέβαιος ότι οι οπαδοί του Τραμπ ε, θέλουν σε ταυτόχρονη βάση να μολύνουν τρεις πλανήτες. Αλλά παρόλα αυτά ας κάνουμε μία μικρή προσπάθεια. Τα μέλη της ΕΝΒΗ, της ΙΤΡΕ και της ΤΡΑΝ προσπάθησαν να εξετάσουν την πρόταση αυτή από την προοπτική την οποία είχαμε ήδη θέσει. Θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι ο τομέας των μεταφορών είναι σημαντικός τομέας για τις εκπομπές και θα πρέπει να ελεγχθεί μέσα από συνθετικές πολιτικές και για την λειτουργία μεγάλων μηχανών και για μικρές μονάδες. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ακριβώς τι έγινε και με την περίπτωση έμεις θα πρέπει να έχουμε μια ικανοποιητική ικανότητα ελέγχου και παρατήρησης και δεν θα πρέπει να αγνοείται γενικότερα το περιβάλλον. Ε, τα δέκα επόμενα χρόνια ίσως φαίνεται ότι είναι λίγο μακριά και γι' αυτό θα πρέπει εμείς να γνωρίζουμε σε τακτική βάση το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, το πού κατευθυνόμεθα και το τι συμβαίνει και δεν θα πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από άλλους ε, ε, τομείς. Μάθαμε πολλά από το παρελθόν και αν πράγματι δεν έχουμε ξεκάθαρους κανόνες, εάν δεν έχουμε σωστή παρακολούθηση και έλεγχο, τότε φοβάμαι ότι θα αποτύχουμε. Είναι σαφές ότι θα υπάρχουν πάντα αυτοί οι οποίοι θα κάνουν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν. Και ταυτόχρονα θα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι συστηματικά δεν κάνουν τίποτα. Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να έχουμε στόχους και ρεαλιστικούς και φιλόδοξους. Merci, Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Ελπίζω όλη η Επιτροπή να συμμερίζεται το στόχο σα για τη διάσωση του περιβάλλοντος. Λοιπόν, και την υποβολή ε, τροπολογιών μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Στις 12 μάλλον το μεσημέρι. Ωραία, α συνεχίσουμε τώρα. με την έκθεση του κυρίου Τέιλορ. Προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσει προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κύριε Σίγητα, έχετε το λόγο. Και μετά θα περάσουμε στους σκιώδες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι έτσι πολύ ε, ελκυστικός ο τίτλος, έτσι δεν λέτε κι εσείς. Ο Ντάβο ήταν ε, ε, εισηγητή ε, στο παρελθόν για αυτό το φάκελο, όμω έχει αποχωρήσει. Επομένω, επειδή δεν έχω κάνει και πολλά για αυτό το φάκελο, εν συντομία θα αναφερθώ στι εργασίε μου. Έχω εργαστεί και στο παρελθόν στον τομέα τη προσβασιμότητα και των μη διακρίσεων σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των επιβατών. Και έτσι γνωρίζω πόσο σημαντική είναι αυτή η νομοθεσία για να διασφαλίσουμε την ε, συνδρομή και ανεξαρτησία, αυτονομία των ε, ατόμων ε, με περιορισμένης κινητικότητας. Και δεν είναι περιπολικό να πει κανείς ότι αυτές οι διατάξεις έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν θεμελιωδώς αλλά και να βελτιώσουν δραματικά τις ζωές των πολιτών μας. Γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό για εμάς το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας να διευρυνθεί στην τροπολογία 8 για να ε, συμπεριλάβουμε και τις ε, πολυτροπικές ε, μεταφορές και με τις δημόσιες συγκοινωνίες όπως το μετρό, τα τρένα, τραμ, τρόλεϊ και λεωφορεία. Εδώ θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και όλες τις πλευρές και στάδια ε, της μετακίνησης από τα μηχανήματα εισιτηρίων μέχρι τα FEE e εισιτήρια. Να κάνουμε ακόμα και διαθετικές αλλαγές ε, στις υποδομές μας. Έχουμε συμπεριλάβει μία σειρά τροπολογιών για να ενσωματώσουμε την κινητικότητα και τον τουρισμό και την πολυτραπική προσβασιμότητα. Για να διασφαλίσουμε ότι η εμπειρία για τους επιβάτες ε, με περιορισμένη κινητικότητα θα ε, βελτιωθεί, θα αυξηθεί και θα είναι προσβάσιμη σε κάθε στάδιο του ταξιδιού της μετακίνησης. Στον, στην τροπολογία 12 έχουμε ένα νέο ορισμό της προσβασιμότητας χωρίς εμπόδια, barrier free. Και θεωρούμε ότι θα πρέπει να μπορεί κανείς να μετακινείται ε, εύκολα και απλά χωρίς ε, να, να αντιμετωπίζει εμπόδια που περιορίζουν την κινητικότητά του. Και τέλος, τριπολογία 5, θίγουμε το ζήτημα της νομοθετικής ε, συνοχής. Και συνιστούμε στην Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει υφιστάμενους κανονισμούς, όπως ο κανονισμός για δικαιώματα των υπερβατών, ως μια βάση νομοθετικών πράξεων για την προσβασιμότητα στις ε, υπηρεσίες ε, μεταφορών και μετακινήσεων. Περιμένω να ακούσω με ενδιαφέρον τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ, κύριε Σιγητά. Ο κύριος Κόχ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το σχέδιο εκθέσεως αποτελεί στέρεα βάση για την περαιτέρω συνεργασία. Ο ορισμός των ατόμων με αναπηρίες καθώς και το θέμα που μάλλον το ζήτημα που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανθρώπους με λειτουργικές αδυναμίες πρέπει να συζητηθούν. Η ιδέα του εισηγητού να περιλάβει και στοιχεία πολυτροπικών μεταφορών είναι πολύ σωστή. Άλλωστε σήμερα το πρωί παρόμοιο ερώτημα έκανα στον Μαλτέζο Υπουργό Μεταφορών, ερώτημα το οποίο δυστυχώς δεν απαντήθηκε. Θεωρώ πάντως ότι η διεύρυνση για να περιλάβει και τον τομέα του τουρισμού είναι μάλλον προβληματική. Εμένα με ενδιαφέρει να δημιουργηθεί μια συνεκτική νομοθεσία που θα είναι σαφή και η οποία δεν θα έρχεται σε σύγκρουση με τις υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει από τη μια μεριά οι κανόνες, οι ρυθμίσεις που ισχύουν για ανθρώπους με ειδικέ ανάγκες σε όλα τα είδη μεταφορών και που εφαρμόζονται εδώ και καιρό να μην υπονομευθούν, αλλά το πολύ να συμπληρωθούν οι κανόνες αυτοί. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να αποκατασταθεί μια σωστή ισορροπία με μεγαλύτερη λήψη υπόψη των αναγκών ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες χωρίς να οδηγηθούμε σε δυσανάλογες επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων. Αναμένω βεβαίω με μεγάλο ενδιαφέρον την ε, συνεργασία με τον εισηγητή και του άλλου συναδέλφου μου. Και ευχαριστώ για την προσοχή που χαρίσατε στα λόγια μου. Η κυρία Σενάλοβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Νομοθετική Πράξη προσβασιμότητα δημοσιεύθηκε πριν από ένα χρόνο και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό βλέπω ότι συμβαίνει σε πολλές επιτροπές. Το συζητήσαμε το θέμα και στην Επιτροπή Εσωτερική Αγοράς που είναι και καθήλυνα αρμόδια. Τώρα σε ό,τι αφορά τη γνωμοδότηση τη επιτροπή μα εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τον εισηγητή ε, για το σχέδιο γνωμοδότησης του. Συμμερίζομαι την ουσία και το πνεύμα ε, της γνωμοδότησης και έτσι δεν έχω πολλά να προσθέσω. βελτίωση των υποδομών, ε, επέκταση του πεδιοφαρμογής στις πολυτροπικές μεταφορές, Όλα αυτά με βρίσκουν σύμφωνοι. Θα υποβάλω κάποιε τροπολογίες σε ό,τι αφορά τα για διαστημικά δεδομένα σε εφαρμογές, σε ό,τι αφορά τις διαδρομές και το προσωπικό των σταθμών. Θα θίξω και τομείς ε, που προς το παρόν δεν καλύπτονται από την νομοθεσία, όπως είναι τα μηχανήματα έκδοσης στηρίων. Δεν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω. Είναι μια πολλά υποσχόμενη γνωμοδότηση και προσβλέπω στη συνεργασία με τον νέο εισηγητή και με οποιονδήποτε άλλο θα ασχοληθεί με αυτό το φάκελο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μπουρμπά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την προσπάθεια την οποία έκανε. το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι οι άνθρωποι με αναπηρίες να μπορέσουν να διασφαλίσουν μια ανεξάρτητη ζωή. Αυτό είναι ο βασικός στόχος αυτών των πρωτοβουλειών. Αυτονομία, ενσωμάτωση κοινωνική, ενσωμάτωση επαγγελματική. Πέρα λοιπόν από όλες τις επιμέρους ρυθμίσεις, συμβάσεις και άρθρα, θα πρέπει να τα ενθυμούμεθα όλα αυτά βέβαια, αλλά να δούμε και ποιες είναι οι υποχρεώσεις τις οποίες δεν έχουμε φέρει πέρας. Θα ήθελα, θα έλεγα να θέσω και ένα θέμα κάπως διαφορετικό. Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο αναπηρία και είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται, είναι μια έννοια η οποία είναι αρνητική. Εγώ θα ήθελα να αλλάξουμε ακριβώς τον κεντρικό μας στόχο η προσαρμογή θα πρέπει να είναι επίσης και μια ευκαιρία για την καινοτομία στην παραγωγή προϊόντων. Είναι κάτι το οποίο θα είναι θετικό για όλους συνεπώς και όχι μόνο για αυτούς οι οποίοι υποφέρουν από ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να τα δούμε τα θέματα αυτά σε επίπεδο επενδύσεων και όχι σε επενδύσεων, σε επίπεδο κόστους μόνο. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να έχουμε τις δυνατότητες επένδυσης για να χρησιμοποιήσουμε τις καινοτομικές διαστάσεις των προϊόντων αυτών και την πρόσβασή του στην αγορά. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει αν θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον όρο πρόσωπα ή πολίτες με λειτουργικούς περιορισμούς. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να ισχύσει, αλλά δεν θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε συλλογικά. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ορίσουμε με πιο θετικό τρόπο την έννοια της αναπηρίας. Πρέπει να βρούμε μία διέξοδο γιατί ο όρος αυτός δημιουργεί κάποιες συγχύσεις. Και φυσικά θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τα άτομα με κινητικούς περιορισμούς και να αναφερθώ και στους όρους τους οποίους έθεσε ε, ο εισηγητής για να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής ε, και σε άλλες μορφές μεταφορά σε αστικούς χώρους, σε αστικές περιοχές. Να υπάρξει δηλαδή ένα γενικότερο πλαίσιο εναρμόνισης. Να συμπεριλάβουμε επίσης και τις τουριστικές δραστηριότητες και τις δυνατότητες να διευκολύνουμε την κινητικότητα αυτό είναι κάτι το οποίο ζητάμε και σε άλλες εκθέσεις. Μιλάμε για την ανάγκη ανάπτυξης του τουρισμού και να ξεπεράσουμε την εποχιακή φύση κτλ. Θα πρέπει να διευκολύνουμε λοιπόν την πρόσβαση σε αυτές τις δραστηριότητες των συγκεκριμένων προσώπων. Και σχετικά τώρα με την τροπολογία 8, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της εφαρμογής σε διάφορα άλλα στάδια θα έλεγα τα οποία εμείς θα πρέπει και αυτά να τα καταστήσουμε ε, προσβάσιμα. Θα πρέπει λοιπόν από την ε, αρχή μέχρι το τέλος μιας δραστηριότητας μετακίνησης να διευκολύνουμε τους ανθρώπους, τις κοινότητες των ανθρώπων οι οποίοι δεν υποφέρουν από αναπηρίες αλλά από μια διαφορετική μορφή κινητικότητας. Αυτό είναι κάτι που τους χαρακτηρίζει. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν κάποιες τροπολογίες και θα συνεργαστούμε με τον εισηγητή έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια ρεαλιστική έκθεση, μια πρακτική έκθεση, μια έκθεση η οποία να λειτουργήσει υπέρ της ανεξάρτητης ζωής. Ευχαριστούμε κύριε Κιλιόναν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η προσβασιμότητα είναι ζωτική σημασία σε, ό,τι αφορά την ισότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε μία ευρεία και καθολική τέτοια προσέγγιση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν αλληλεπικαλύψεις στην νομοθεσία μας. Ήδη έχουμε κάποιες προβλέψεις, για παράδειγμα, στα συνδρομικά δίκτυα. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος να τα μπερδέψουμε, να δημιουργήσουμε ε, αντιφατικές ε, απαιτήσεις και κανόνες στις επιμέρους νομοθετικές πράξεις. Πρέπει να θέσουμε τα θεμέλια για τη διασφάλιση μιας καλύτερης προβασιμότητας για όλους. Ξέρω ότι υπάρχουν οι δήμονες που έχουν έρθει σε επαφή με πολλούς από εμάς. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από τον εισηγητή και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς ακριβώς ε, θα διασφαλίσουμε αυτή την ε, συνεκτική και λογική ε, νομοθεσία για να αποφύγουμε τις αλληλεπικαλύψεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την έκθεση επίσης, την εισηγήτρια δηλαδή. Πάντοτε είναι θετική κάθε προσπάθεια διασφάλισης πρόσβασης σε ανθρώπους με αναπηρίες. Οι χώρες μέλη έχουν διαφορετικές αφιθυρίες. Ας μην το λησμονούμε. Από αλλού ξεκινούν οι διάφορες χώρες, η κάθε μία δηλαδή. Εδώ έχω ορισμένες προτάσεις, προτάσεις βελτιώσεως. Θεωρώ ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε ήδη ρυθμίσεις ειδικέ ανατομέα η TSPRM για τα δικαιώματα των επιβατών. Έχουμε ήδη επιτύχει ορισμένα πράγματα και δεν χρειάζεται, δεν έχουμε κανένα λόγο να, να, να ντρεπόμαστε. Έχουμε επιτύχει λοιπόν πολλά και σημαντικά πράγματα. Τώρα, χρειάζεται βέβαια και σόφρον προσέγγιση και να εργαστούμε με καλή πρόθεση αλλά και με καλά αποτελέσματα. Δηλαδή, να μην λησμονούμε την αναλογικότητα. Αν έχω καταλάβει καλά, κάθε αυτόματο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων θα πρέπει να έχει εξοπλιστεί εκ νέου, ας πούμε έτσι, να έχει εξυγχρονιστεί μέσα σε έξι χρόνια. Επιτυχάνουμε έτσι το σκοπό μας, ερωτώ. Ή ίσως πάμε εκεί να δαπανίσουμε χρήματα με άσκοπο τρόπο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλού. Διότι έχουμε τα εφή e τηλέφωνα με πάρα πολύ ψηλούς αριθμούς ανθρώπων οι οποίοι κλείνουν τα εισιτήριά τους μέσω των εφιών τηλεφώνων τους. Ψηφιοποίηση, διαδίκτυο κλπ. Ε, εξέτασα τον γερμανικό τύπο και έπεσα σε διαφήμιση των γερμανικών σιδηροδρόμων που από τον Ιανουάριο μέχρι, το Δεκέμ, μέχρι τον Σεπτέμβριο μάλλον, σε εννέα μήνες, μέσα στο 2016, επόλυσε 6,9 εκατομμύρια εισιτήρια. Και η τάση είναι αυξητική. Ως άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος πάντοτε ήμουν και είμαι υπέρ της αύξησης της κινητικότητας, της διευκόλυνσης της κινητικότητας όλων, ούτως ή άλλως, αλλά και ιδίως αυτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κίνηση, διερωτώμε αν όντως πετυχαίνουμε τον σκοπό μας βάζοντας δε και καλά ένα στόχο που θα πρέπει να επιτευχθεί οπωσδήποτε μέσα σε έξι χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να το επανεξετάσουμε. Ένα άλλο θέμα είναι, κατά τη γνώμη μου, αν πάλι άκουσα καλά, υποτίθεται θα γίνει διάκριση ανάμεσα σε ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών και στο δημόσιο που παρέχει υπηρεσίες. Εδώ κάπως με ενοχλεί αυτό από άποψη δικαιοσύνης. Γιατί σε αυτό το σημείο πάμε να επιβαρύνουμε λιγότερο τους ιδιώτες και το δημόσιο, το οποίο ούτως ή άλλως δραστηριοποιείται για να προσφέρει καθολικές υπηρεσίες. Γιατί προβαίνουμε σε αυτή τη διάκριση. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον εισηγητή. Γιατί δεν είναι δυνατόν ένα πρόσωπο με περιορισμένη κινητικότητα, εάν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχουν ιδιώτες, να είναι υποχρεωμένο να παραιτηθεί από κάποια διευκόλυνση, ενώ για το δημόσιο να μην ισχύει αυτό, να είναι υποχρεωμένο ότι την παράσχει. Τέλος. Εξετάζοντας το σύνολο των διατυπώσεων εννοούν εδώ οι συγγραφείς τις υπηρεσίες ή εκτός των υπηρεσιών και το σύνολο των υποδομών. Γιατί πάλι εδώ η διατύπωση για μένα τουλάχιστον δεν είναι πολύ ξεκάθαρη. Μιλεί για internal entities, εσωτερικές οντότητες, όπου εγώ διαρωτώ θα ισχύει ας πούμε και για τα διοικητικά κτίρια των παρόχων των υπηρεσιών. Διότι αυτό για μένα δεν είναι δικής μας αρμοδιότητας, είναι εθνικής αρμοδιότητας. Άλλο λοιπόν παροχή υπηρεσιών στις υποδομές και άλλο τούτο εδώ. Ας το επανεξετάσουμε λοιπόν και αυτό προσεκτικά. Εδώ ο συγητής προχωρεί ακόμη περισσότερο. Μιλεί και για την υγεία Εγώ επαγγελματικά προέρχομαι από το τομέα τη υγεία, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι παρόλα αυτά τι εννοεί. Και για νέε υπηρεσίε κινητικότητα, όπου πάλι δεν αντιλαμβάνομαι τι ακριβώ εννοεί. Πρόκειται για μια καταρχήν καλή έκθεση που πρέπει όμω να βελτιωθεί. Και βεβαίω πάντοτε με τρόπο εύλογο. Όπω είπα, να μην κατασπαταληθούν χρήματα που μπορεί να πιάσουν τόπο κάπου αλλού. Βήμ, εσύ σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αντλώ έμπνευση από τον συνάδελφό μου τον Ισμαήλ και θα ήθελα να ρωτήσω τον Κιθ Τέιλορ κυρίως σε ό,τι αφορά την... Να του ζητήσω μάλλον να συμπεριλάβει στοιχεία που άπτονται της υλοποίησης της κείμενης νομοθεσίας. Ε, στο ΕΛΚ είχαμε έναν ε, φοιτητή από τη Μολδαβία με αναπηρία ε, που έρχεται στο κοινοβούλιο Ήθελε να έρθει λοιπόν, αλλά ο οδηγός δεν μπορούσε να κατεβάσει η ράμπα για να ανέβει με το καροτσάκι ο φοιτητής. Επομένω, το σημαντικό είναι να αξιοποιήσουμε και να εφαρμόζουμε πιο αποτελεσματικά τι ε, υφιστάμενε δυνατότητε. Βέβαια, πάντα θα πρέπει, θα υπάρχει μάλλον θα πρέπει, θα, υπάρχουν αδυναμίε, αλλά α μην επικεντρωνόμαστε πάντα στην ε, διαμόρφωση νέων δομών, α σταθούμε ε, στην αξιοποίηση των υφιστάμενων. Αυτό θα ήθελα να το τονίσουμε και πάλι. Ευχαριστούμε κύριε Βαντερκάμπ. Να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τρία λεπτά. Εμμανουέλ Γκράνζ. Είναι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Εμμανουέλ ε, επικεφαλή τη ε, μονάδα μου δεν μπορούσε να έρθει εδώ. Ονομάζομαι Είμαι Απλαθένθια. Είμαι επικεφαλή εμπειρογνώμων για ε, ζητήματα προσβασιμότητα στη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή αυτή γνωμοδότηση με την οποία στηρίζει την πρότασή μας ε, που βασίζεται στην ενιαία αγορά αλλά στην γνωμοδότησή του έχει συμπεριλάβει και στοιχεία βελτίωσης σε ό,τι αφορά την ε, κινητικότητα και προσβασιμότητα στις υπηρεσίες μεταφοράς των ατόμων με αναπηρίες. Έχουμε δει το, τη σημασία που αποδίδει στην ανάγκη βελτίωση της προσβασιμότητας ε, σε αυτές τις υπηρεσίες, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογή, όπως οι αστικές συγκοινωνίες, ε, πολυτροπικές συγκοινωνίες και ούτε καθεξής. Και σημειώνουμε για την πρόταση του εισηγητή βελτίωσης ε, των υποδομών. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι υπάρχει ένα έτοιμα στην γνωμοδότηση ε, να αλλάξουν οι φυστάμενοι κανονισμοί και εμείς, ε, εμάς μας προβληματοποιεί, προβληματίζει αυτό το σχόλιο, γιατί δεν υπάρχουν προθέσεις και σχεδιασμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τροποποίηση των κανονισμών για να συμπεριληφθεί η προσβασιμότητα. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και ε, για την ε, ε, αστική κινητικότητα, την αηφόρα αστική κινητικότητα. Η ευθυγράμμιση με τους ισχύοντες κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία είναι πολύ σημαντική για εμάς είμαστε πεπισμένοι ότι η συμπληρωματικότητα των δύο προτάσεων, δηλαδή της νομοθετικής πράξης προσβασιμότητας με ε, τον ισχύοντα κανονισμό ε, για τα δικαιώματα των επιβατών, είναι κάτι το οποίο θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό. Βέβαια, αυτή η πρόταση ε, εστιάζει περισσότερο την προσοχή της στην κινητικότητα, στην προσβασιμότητα, ενώ οι υπόλοιπε προτάσεις στην αρρωγή. Ε, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η έννοια των ατόμων με ε, κινητικούς περιορισμούς έχει ως στόχο να καλύψει όλα τα άτομα που μπορεί ενδεχομένως να μην αναγνωρίζονται επισήμως ως άτομα με αναπηρία, αλλά παρουσιάζουν ε, κάποιες ε, ανάγκες ως προς την προσβασιμότητα. Συνοχή λοιπόν και συμπληρωματικότητα με την ε, νομοθεσία που αναφέρθηκε προηγουμένω και στα σιδηροδρομικά δίκτυα και εν κατακλείδη να πω ότι η πρόταση δεν επιβάλλει την εγκατάσταση ε, μηχανημάτων εκδοση ε, εισιτηρίων, ούτε επιβάλλει την χρήση smartphone. Απλώς λέει ότι όταν χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι προσβάσιμα. Δίνει λοιπόν χώρο για την ε, εξέλιξη για την καινοτομία και αυτό προκύπτει και από την πρόταση. Ευχαριστώ. Ο εισηγητή, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Κύριε Τέλερ, μισό λεπτό. Ευχαριστούμε την Επιτροπή Έχετε το λόγο. Βλέπουμε τον ενθουσιασμό σας ε, για αυτή τη γνωμοδότηση. Το μικρόφωνο του συγητή δεν είναι ανοιχτό. Ενδιαφέρουσες ε, οι παρατηρήσεις σας. Θα τις ε, σκεφτώ προσεκτικά. Επειδή μόλις τώρα έχω αναλάβει τον ρόλο του εισηγητή, μπορεί να καταφέρουμε να ε, διοργανώσουμε μία ε, συνάντηση των σκιωδών για να εξετάσουμε πιθανές συμβιβαστικέ τροπολογίες. Προς το παρόν θα τα εξετάσουμε προσοχή όλα αυτά που είπατε. Μου άρεσαν κάποιες... Ε, μου προκάλεσαν εντύπωση κάποιες ιδέες όπως η αποφυγή των αλληλεπικαλύψεων πώς θα βελτιώσουμε τη ζωή, την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρίες, αλλά και οι προτάσεις προς την καινοτομία. Πολύ καλά όλα αυτά. Όμως επειδή και εγώ κατά καιρού χρησιμοποιώ τον αναπηρικό καροτσάκι, να σας πω ότι αν θέλω να βγω από εδώ μέσα και θέλω να πάω σε ένα καφέ ή ένα εστιατόριο, θα έχω πραγματικό πρόβλημα. Θα δυσκολευτώ πάρα πολύ να βρω ε, κτίριο, μέρος που να μην ε, πρέπει να ανέβω σκαλιά. Πραγματικά είναι αδύνατο να βρω ε, καφέ με ε, την τουαλέτα στο ισόγειο. Συνήθως είναι σε όροφο ή στο υπόγειο με μία ε, σκάλα αρκετά δύσβατη κιόλα. Επομένω, πρέπει να ε, δώσουμε την απαραίτητη σημασία και στα βασικά. Πέραν της αξιοποίησης ε, όλων των ε, ε, τεχνολογιών που έχουμε στη διάθεσή μας για να καλύψουμε τις ανάγκες αυτών των ατόμων με αναπηρίες και για να τους επιτρέψουμε να ζήσουν τη ζωή τους στα έπακρον. Ευχαριστούμε κύριε Τέιλορ. Συνεχίζουμε. Sur le rapport de Monsieur Taylor. Λοιπόν, για την έκθεση Taylor υποβάλλεται τροπολογίες μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Continuons avec l'examen, la présentation par la Commission. Ας συνεχίσουμε τώρα σε ό,τι αφορά την παρουσίαση από την Επιτροπή των της Υπράξεων σχετικά με τις κατευθύνες γραμμές των TNT. Έχει 10 λεπτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ε, παρουσιάσει αυτές τις ε, κατευθυντήριες γραμμές, ε, συγγνώμη, της κατευθυντήρες πράξης βάσει του άρθρου 49.4 και 49.6. Το 49.4 αφορά την ε, προσαρμογή ε, των χαρτών και της γενικής εφαρμογής μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο. Σας έχει έρθει η ενημέρωση από το newsletter της Επιτροπολογίας αυτή τη στιγμή πριν τεθεί σε ισχύ μεταφέρεται το σχέδιο καταξιδίου της πράξης προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και η δεύτερη καταξιδίου πράξη, πράξης, 49.6 άρθρο, αφορά την ε, συμπερίληψη των ενδεικτικών χαρτών των γειτονικών χωρών που έχουν τεθεί υπό διαπραγμάτευση και θα μας παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι συμβαίνει και υπενθυμίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό που η δική μας Επιτροπή ε, παρακολουθεί εκ του τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί τις ε, εξουσίες τις οποίες ε, τις έχει παραχωρήσει το Κοινοβούλιο. Για ένα από τα πιο σημαντικά νομοθετικά μέτρα σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές μεταφορές και σας καλώ συνάδελφοι να Διαβάστε με μεγάλη προσοχή τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α δώσουμε τώρα το λόγο στο Φρέντερικ Βελσινή από τη Γενική Διεύθυνση MOVE της Ευρωπαϊκή Επιτροπής και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στον ε, εισηγητή κύριο Μάρκος Πίπερ που δεν βλέπω προς το παρόν βέβαια εδώ και ο Ισμαήλ Ερτούκ θα πάρει το λόγο στη συνέχεια. και μετά θα δώσουμε το λόγο και στους συντονιστέ και στα μέλη που επιθυμούν να πάρουν το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ που ζητήσατε την Επιτροπή να παρουσιάσει αυτές τις δύο κατεξουσιοδότηση πράξεις. Ήδη θέσατε το πεδίο εφαρμογής αυτών των δύο πράξεων σε προκαταρκτικό επίπεδο θα ήθελα να χαιρετήσω καταρχάς την συνεργασία που υπήρξε ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Το Κοινοβούλιο ενημερώθηκε τακτικά. Η πρώτη κατεξουδότηση πράξη αναφέρεται στην επικαιροποίηση και την τακτική παρακολούθηση του δικτύου RTT. E Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σε ισχύ τον κανονισμό ατήτη έχουν γίνει σημαντικά βήματα καρπός της κοινή προσπάθειας των τριών θεσμικών οργάνων έτσι ώστε να προχωρεί το σύστημά μας στην Ευρώπη και η δεύτερη κατεξουσιοδότηση πράξη αφορά στις σχέσεις μας με τις γειτονικές χώρες. Αν μου επιτρέπετε τώρα θα συνεχίσω στα αγγλικά. Πριν παρουσιάσω κάθε μία από τις κατεξιοδότηση πράξεις, να υπογραμμίζω ότι και στις δύο περιπτώσεις δεν συνδέονται οι δύο περιπτώσεις ε, με την χρηματοδότηση υποδομών, με τη χρηματοδότηση γενικότερα, όπως επίσης και με τον καθορισμό των διαδρόμων, όπως επίσης ε, και των Lifeline Corridors. Να ξεκινήσω λοιπόν με την πρώτη κατεξουσιοδότηση πράξη για τη στατιστική ενημέρωση των TNT, επικαιροποίηση μάλλον των TNT. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί από κοντά την, των τεχνικών παραμέτρων και το άρθρο 49.4 δίνει την δυνατότητα υιοθέτησης κατεξουσιοδότηση πράξεων έτσι ώστε να ενημερώνονται τα παραρτήματα 1 και 2 και να λαμβάνονται υπόψη πιθανές αλλαγές οι οποίες προέρχονται από τα ποσοτικά όρια τα οποία έχουν καθοριστεί ε, για την διάκριση των ε, συστατικών υποδομών στο σύνολο των δικτύων. Να σας ενημερώσω για τη διαδικασία που ακολουθήσαμε. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία αυτή επικαιροποίηση στις 30 Σεπτεμβρίου του 2015 σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές επί τη βάση δελτίων τα οποία περιέχονται στο σύστημα των TNT. Την παρουσία εκπροσώπων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις ομάδες εμπειρογνωμόνων επίσης ε, έγιναν συναντήσεις, μία στις 9 Δεκεμβρίου του 2015 και στις 16 Μαρτίου και 16 ε, ε, Σεπτεμβρίου του 2016. και 7 Δεκεμβρίου έγινε δεκτή η κατεξουσιοδότηση πράξη η οποία σας απεστάλλει. Οι προτάσεις οι οποίες γίνονται αναφέρονται σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι ρυθμίσεις ε, στους χάρτες έτσι ώστε να ε, αντιπροσωπεύουν την πρόοδο που έχει γίνει στα δίκτυα. Δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στο σύνολο των δίκτυων αυτών όταν τα ποσοτικά επίπεδα έχουν ξεπεραστεί. Αυτό αναφέρεται και στην εσωτερική ναυτιπλοεία, στην ακτοπλοεία και στις πολυτροπικές, ε, ε, ε, ε στις πολυτροπικές μεταφορές. Όλες αυτές οι υποδομές λοιπόν παρακολουθούνται σύμφωνα με τις στατιστικές τις οποίες μας παρέχει η Eurostat. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 250 αιτήσει τροποποίησης, 235 μπορούσαν να γίνουν δεκτές. Απορρίψαμε 15 αιτήσει και ο λόγος για τους οποίους τις απορρίψαμε ήταν διαφορετικές. Υπήρχαν αιτήματα εκτός του πεδίου εφαρμογής υπήρχαν αλλαγές στο κομβικό, στο κεντρικό δίκτυο και η προσπάθεια αυτή δεν ασχολείται με το κεντρικό δίκτυο, αναφέρεται μόνο στα επιμέρους δίκτυα. Άλλοι λόγοι απόρριψης είχαν σχέση με το ανώτατο όριο το οποίο δεν είχε επιτευχθεί, όπως επίσης και με την συνένωση επιμέρους στόχων. Από τις 235 οι 211 αφορούσαν προσαρμογές σε προόδους που είχαν γίνει σε οδικά δίκτυα, σε οδρομικά δίκτυα και ε, εσωτερική ναυσιπλοεία στο συνολικό δίκτυο. Ε, λιμένες εσωτερικής ε, ναυσιπλοείας, εμπορευματικές μεταφορές και ένα αεροπόριο αεροδρόμιο, συγγνώμη. Ε, ταυτόχρονα σκοπεύουμε στο μέλλον η διαδικασία αυτή να μην γίνεται σε αιτήσια βάση, αλλά να δύο ή τρία χρόνια σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Τώρα να μου επιτρέψετε να έλθω στη δεύτερη κατεξουσιοδότηση πράξη, την επέκταση δηλαδή του δικτύου TNT. Ε, το παράρτημα 3 του TNT, του κανονισμού TNT, όταν υιοθετήθηκε το 2013, περιελάμβανε ήδη ορισμένους ενδεικτικούς χάρτες για τις γειτονικές χώρες. Οι γειτονικές χώρες, οι χώρες γειτονίας μάλλον, οι οποίες έχουν τη στενότερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν ε, ε, και Ελβετία. Υπήρξαν λοιπόν ορισμένοι ενδεικτικοί χάρτες και για την Τουρκία και για τα Δυτικά Βαλκάνια. Το άρθρο 49.6 του κανονισμού προβλέπει την δυνατότητα να υιοθετηθούν κατ' εξουσιοδότηση πράξη προσαρμογής αυτός, αυτών των ενδεικτικών χαρτών, γεωγραφικών χαρτών, στα πλαίσια της συμφωνίας βέβαια ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες γειτονίας. Τα προηγούμενα χρόνια έγινε σημαντική πρόοδος με στόχο την ενίσχυση ακριβώς της συνεργασίας αυτής. Τα δίκτυα αυτά καθορίστηκαν και για τα Δυτικά Βαλκάνια και για την Τουρκία και για τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία, Γεωργία, Αρμενία, Ουκρανία και Ρωσία. Ενθυμίστε ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε περάσει μια κατεξουσιοδότηση πράξη ε, για τα Δυτικά Βαλκάνια. Τώρα προτείνουμε να γίνει ένα βήμα επιπλέον και να ορίσουμε επίσης και τα κομβικά δίκτυα και στην Τουρκία και στις χώρες ανατολικής γειτονίας. Η συμφωνία υψηλού επίπεδου ανάμεσα στην Ένωση και τις συγκεκριμένες χώρες επετέφθη στις ε, 21 Ιουνίου του 2016 στο Ρότερνταμ στα πλαίσια ε, των, της ημερίδας για τα 10 που είχαμε εκεί και υπήρξε συμφωνία με τους νέους ενδεικτικούς χάρτες οι οποίοι θα προταθούν στην κατεξουσιοδότηση πράξη. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές, την παρουσία εκπροσώπων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ομάδων εμπειρογνωμόνων που συνεδρίασαν το Δεκέμβριο του 2015, το Μάρτιο, το Σεπτέμβριο και το Δεκέμβριο του 2016. Συνεπώς λοιπόν ο κανονισμός αυτός αναμένεται να υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του μήνα, στις 31 μάλλον Ιανουαρίου και θα αποσταλεί τότε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βασικός μας στόχος είναι να επιτρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να στοχεύσει καλύτερα τη συνεργασία και σε επίπεδο δημοσιονομικής στήριξης των γειτόνων, μια προσπάθεια η οποία δεν δημιουργεί νέα δικαιώματα οικονομικά για τις χώρες αυτές, αλλά η βασική μας ιδέα είναι να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στις κοινέ προτεραιότητες και να διασφαλίσουμε με τον τρόπο αυτό ότι οι γειτονικές χώρες εφαρμόζουν τα ίδια standards, τα ίδια επίπεδα δηλαδή για την ανάπτυξη των υποδομών. Να πω ότι μια αντίστοιχη προσπάθεια γίνεται και με τις μεσογειακές χώρες. Δεν έχει υπάρξει ακόμα μια συμφωνία στο Ρότερνταμ τουλάχιστον στις ημερίδες T με τις χώρες αυτές αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα κοινό ορισμό των δικτύων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για να δώσω απαντήσεις εφόσον το επιθυμείτε. Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε της Επιτροπής για την πλήρη απάντηση. Αλλά μπορείτε να μιλείτε για γαλλικά εφόσον το επιθυμείτε. Εσεί, κύριε Σιγητά, κύριε Ισμαήλ ε, Ερτουκ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έχω πει πάντοτε και θα το επαναλάβω. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι ίσω, παράλληλα και με το πρόγραμμα Έρασμος ΣΥΝ αυτά εδώ τα Ευρωπαϊκά δίκτυα είναι το καλύτερο πράγμα που έχει να επιδείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους και στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όλες και όλους που έχουν συνεργαστεί για το ίδιο αυτό, για τον ίδιο αυτό σκοπό. Στην τελευταία περίοδο χαράξαμε τις βασικές γραμμές των δικτύων και είχαμε λίγο το όραμα του μέλλοντος 2021 να κάνουμε αναθεώρηση. Ακούγοντας τώρα την απάντηση της Επιτροπής, αντιλαμβάνομαι ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα και μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε συνεργασία με τις γειτονικέ μας χώρες. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με βοήθεια αυτών των υποδομών και των σχετικών έργων έχει στα χέρια και έναν γεωπολιτικό μοχλό που συχνά δεν λαμβάνουμε υπόψη. Μιλούμε για μεγάλους πολιτικούς στόχους, ενώ με αυτά τα μέτρα υποδομών, ξαναλέγω, έχουμε στα χέρια μας ένα γεωπολιτικό εργαλείο που θα πρέπει να μας καθιστά υπερήφανους. Το ερώτημά μου είναι, εκτός τώρα από τα πολλά λόγια επένων που ήδη εξέφρασα, Απευθύνομαι τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαρωτώ με κατά πόσον προετοιμάζει την αναθεώρηση των διευρωπαϊκών δικτύων και αν σκοπεύει να αρχίσει την προσπάθεια αυτή. Τι, πώς μπορεί να τα στρέψει στο μέλλον, που εκτός από όλα αυτά τα θετικά στοιχεία υπάρχουν και αρνητικά. Έχουν περάσει τρία-τέσσερα χρόνια. Νομίζω θα πρέπει να είμαστε πλέον σε θέση να μπορέσουμε να κάνουμε τουλάχιστον μια δήλωση σχετικά. Ευχαριστώ κύριε Τιούγκ. Ο κύριος Βάντερ Κάμπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, όντω δεν είναι εδώ μαζί μα ο Μάρκο Πίπερ, συνεισηγητή, αλλά θα δούμε εσωτερικά τι ακριβώ συνέβη, γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι πολύ παλιό ο φάκελο και πεπειραμένα ε, μέλη όπω ο Έρτουφ και ο Πίπερ πρέπει να ασχολούνται με αυτό το φάκελο. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ο διάβολο κρύβεται στι λεπτομέρειε. Αυτό είναι το δεύτερο που ήθελα να φέρω. Προηγουμένως ε, εξετάσαμε ένα ε, θέμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό με τεράστιες προεκτάσεις, όπως είναι και αυτό τώρα με τα δίκτυα, ε, τα δίκτυα μεταφορών. Και αύριο το πρωί θα εξετάσουμε μία έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για τις επενδύσεις στους λιμένες. Και θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια τέτοια έκθεση επηρεάζει τις επενδύσεις ε, τεντή Και ο κύριος Σέρτουκ το ανέφερε ότι ε, τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών είναι μια τεράστια επιτυχία, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί που ακριβώς επενδύουμε. Κανείς δεν ωφελείται από άδεια αεροδρόμια. Όπως είπε και ο κύριος Κράμερ, για όλα αυτά τα περιφερειακά αεροδρόμια που έχουμε, τα οποία δεν είναι εκμεταλλεύσιμα. Επομένω, ε, πώ έχουν τα πράγματα ω προ αυτέ τι επενδύσει. Μετά, ο συνάδελφο Μαρία Μαρινέσκου ε, μου ανέφερε να σας, και ζήτησε να σας πω ότι χαιρόμαστε που οι καταξιδότηση πράξη συνάδουν πλέον με τις ε, αποκαλούμενες κατευθύνες γραμμές TNT. Αυτό είναι θετικό και δεύτερον είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που το μικρό αυτό κομμάτι που έλειπε μεταξύ Ρουμανίας και Βουλγαρίας και είχε αναφερθεί στο παρελθόν στην Επιτροπή Μεταφορών, έχει λυθεί πλέον το πρόβλημα. Αυτό δηλαδή το ε, τμήμα των 10 χιλιόμετρων που έχει καλυφθεί πλέον. Και ε, σας ευχαριστώ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Αιάρα Σέντερ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δύο κατεξουσιοδότηση πράξεις, οι οποίες πράγματι έχουν σημασία και έπρεπε να γίνουν οι διαρρυθμίσεις αυτές, μιας και πρόκειται για χάρτες. Είναι κάτι το ιδιαίτερο χρήσιμο για τους εκπροσώπους, τους περιφερειακούς, τους τοπικούς. Και αν δεν είναι σωστοί δημιουργούν πάρα πολλά θέματα στους ίδιους ανθρώπους. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να ε, διορθώσει κανείς τους χάρτες αυτούς σε επίπεδο λεπτομέρειας, αλλά νομίζω ότι έχει σημασία να δούμε ακριβώς και τι αλλαγές έχουν γίνει και στον τομέα των σιδηροδρομικών γραμμών. Έχουμε μία εδώ που ξεκινάει από το Βαγιαλοδρίδι προς το Σαταντέρ και από το Βαγιαδολίδια τη Βικτόρια. Εδώ δεν μπορούμε να δούμε, δεν μπορούμε να καταλαβήσουμε αν πράγματι ε, πρόκειται για γραμμές υψηλής ταχύτητας ή κάτι άλλο. Δεν βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται. Δεν είναι ιδιαίτερα αναγνώσιμοι οι συγκεκριμένοι χάρτες. Ξέρω ότι το θέμα δεν είναι θέμα το οποίο μπορεί η Επιτροπή να δει, αλλά σε επίπεδο σχεδιασμού του χάρτη υπάρχει εδώ ένα θέμα. Και στο νότο τώρα έχουμε τη γραμμή ανάμεσα στην Αλμερία και τη Γρανάδα. Και εδώ είναι μια γραμμή η οποία έχει αρκετά μεγάλη σημασία. Όχι τόσο στο χάρτη, αλλά στην έκθεση του κυρίου Μπρέινχορστ μπορεί να δημιουργήσει κάποια θέματα, γιατί οι τοπικές αρχές και οι πολίτες άσκησαν κριτική στο ότι δεν είχαν υπάρξει λοιπόν επενδύσεις που απαιτούνται. Λοιπόν, στο πρώτο θέμα είναι θέμα χάρτη, τεχνικής, αν θέλετε, χαρτογραφικής. Και στο δεύτερο να πω ότι όταν οι, συγητές, οι συντονιστές παρουσίαζαν τις εκθέσεις τους υπήρχε μια τέτοια πρόταση, μια παρουσίαση και στη δική μας Επιτροπή στο παρελθόν αλλά τώρα βλέπουμε ότι έχουν δημοσιευθεί χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς ε, ε, ποιοι είναι υπεύθυνοι και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα υποστούν, αν θέλετε, τις αλλαγές αυτές, όπως οι τοπικές αρχές, οι δήμαρχοι και ο τοπικός πληθυσμός γενικότερα. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα πλέον θα πρέπει να ζητήσουμε πλέον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά τα οποία έκανε στο παρελθόν και να πούμε θα πρέπει να υπάρχει σωστή ενημέρωση σε σχέση με την επικαιροποίηση για την κατάσταση, της αλλαγές που έχουν εντωμεταξύ συμβεί και να υπάρχει μια κάποια προειδοποίηση, εν περιπτώσει, για τις αλλαγές αυτές. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Σενάλοβα, για την παρουσίαση του θέματος. Και έχω και μία πιο εξειδικευμένη ερώτηση. στο παράρτημα 1 του 1738 δεν αναφέρεται η γραμμή Μπρνό-Φερόφ. Στην προηγούμενη ωστόσο εκδοχή του κανονισμού περιλαμβανόταν στο παράρτημα 1 του 1433. Διαρωτώ με εάν πρόκειται για αυλευσία ή εάν πρόκειται για εσκεμμένη παράληψη. Και αν όντω έγινε εσκεμμένα η παράληψη αυτή, ρωτήσατε καθόλου την τσεχική δημοκρατία τι γνώμη έχει. Διότι το άρθρο 49 γάμα λέει ότι οι διαδρομές μπορούν να μεταβληθούν μόνο μέσω επίσημης διαδικασίας έγκρισης έργων. Ευχαριστώ. Πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Κύριε Θέλω να κάνω μια συγκεκριμένη αναφορά, να πω ότι η νομοθεσία σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα να γίνονται διάδρομοι μεταφορός ε, εμπορευμάτων επί τη βάση διακρατικών συμφώνιων. Και αναφέρομαι στον διάδρομο Άμπερ, στον διάδρομο 11, και την ε, προσπάθεια ένταξης του διαδρόμου αυτού στα TNT. Πώς ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προωθήσει τη συνεργασία ανάμεσα στους λιμένες της Βαλτικής και τους λιμένες της Αδριατικής. Ενώ ε, ε, έχουμε να κάνουμε με δύο λιμένες σχετικά κοντά ο ένας τον άλλο, σημαντικούς για την περιοχή της Αδριατικής, την Τευγέστη και το Κάπο και να δούμε ακριβώς πώς τα τέντη συνδέονται με τους λιμένες και με άλλους ιδεοδρομικούς διαδρόμους. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν αν θα μπορούσαμε να έχουμε και μία συνάντηση με την Επιτροπή μας σαν και αυτή που είχαμε στις 5 Δεκεμβρίου όταν είχαν ληφθεί οι αποφάσεις για τους επιπλέον διαδρόμους να υπάρξει δηλαδή καλύτερο συντονισμός ανάμεσα στις δραστηριότητές μας έτσι ώστε να γνωρίζουμε εγκαίρως ε, τις αποφάσεις αυτές οι οποίες πολλές φορές χρήζουν συζήτηση σε βάθος. Ευχαριστώ πολύ. Κράμερ. Τελευταία παρέμβαση. Είπε προηγουμένως ο Βιμ Φαντεκάμπ Κάμπ για την έκθεση για τα περιφερειακά αεροδρόμια. Πραγματική καταστροφή. Τα χρήματα, τα ευρωπαϊκά χρήματα που επενδύθηκαν εκεί δεν είχαν σχεδόν κανένα αποτέλεσμα. Όλα τα νούμερα που είχαν δοθεί δεν επετεύχθησαν. Ήταν καθαρή κατασπατάληση χρήματος. Αύριο θα ακούσουμε έκθεση για τα λιμάνια. Μήπως νομίζω ότι εκεί θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Άλλη καταστροφή από εκεί. τρία λιμάνια σε απόσταση 5-10 χιλιόμετρων μεταξύ τους επιδοτούνται με ευρωπαϊκά χρήματα και το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Μα τι τις κάνετε τις εκθέσεις αυτές μου λέτε. Τι επιπτώσεις έχουν. Απλά συνεχίζετε. Ποιες είναι οι επιπτώσεις που, πια είναι τα διδάγματα που αντλείται από αυτά. Διότι οι χώρε μέλη βεβαίω χαίρονται που λαμβάνουν τα χρήματα αυτά. Χαίρεται η οικοδομική ε, βιομηχανία, η οικοδομή, χαίρεται ο οικοδομικός κράτος και οι τράπεζες. Αλλά το αποτέλεσμα σας ξαναλέω είναι μηδέν. Στο μέλλον επιθυμείτε, δηλαδή έχετε σκοπό να ξανακάνετε τα ίδια λάθη. Στο σχολείο λένε από τα λάθη γίνεται κανείς σοφότερος. Αλλά εδώ δεν μου φαίνεται να συμβαίνει αυτό σε εσά. Δεύτερο, μπορεί να εγγυηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η διαδικασία της επιτροπολογίας θα σέβεται και τα κριτήρια. Κριτήρια σημαίνει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ελαχιστοποίηση των εξωτερικών στοιχείων κόστους και οι cross-border connections, οι διαμεθοριακές διασυνδέσεις. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα στο οποίο αναφέρομαι. Είχαμε τα 110 εκατομμύρια, τα ανέφερα σήμερα το πρωί, πολύ σημαντικά ποιες είναι οι συνέπειες να πιεστούν οι χώρες μέλη να μην σκέφτονται μόνο τα μεγάλα έργα αυτοπροβολής τους, αλλά και τα μικρότερα διαμεθοριακά έργα, τα οποία δεν ενδιαφέρουν τους υπουργού καθόλου, σαν να μην υπάρχει καν η Ενωμένη ΕΕ. Δεύτερο, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν για παράδειγμα η οδηγία UVP δεν εφαρμόζεται. Μου ελέγχθη ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, φαίνεται πως είναι και οι Δήμων περί την πολιτική μεταφορών αλλά και τη χρηματοδοτική πολιτική, τους είπε στους Τσέχους για την κατασκευή 10 δρόμων δεν χρειάζεται να λάβετε υπόψη σας καν την οδηγία UVP. Είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Πού ζούμε, σε τι κόσμο ζούμε. Μπορεί να βγει ο πρόεδρος Επιτροπής και να πει απλώς παραβιάζω τα νομοθετικά κείμενα. Τι κάνετε ως Επιτροπή. Τα ελέγχετε αυτά τα πράγματα. Δεν έχω ακούσει τίποτα σχετικά. Τα έμαθα μόνο από τους ενδιαφερόμενους Τσέχους. Τρίτο, κάτι εξουσιοδότης είναι πράξεις. Είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι σε αυτές. Περιλαμβάνονται μεν στην συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά η εμπειρία μου εδώ στο Κοινοβούλιο είναι ότι Κομισιόν και Συμβούλιο κάνουν τα πάντα για να τις θέσουν στην πράξη εκτός ισχύω. Εάν τα, τα διευρωπαϊκά δίκτυα που έχουν εγκριθεί από όλους εδώ εμάς εφόσον διευρυνθούν, είναι απλά δηλαδή τι είναι, τεχνικό θέμα, επομένως δεν μας ρωτάτε. Γιατί όχι, προδιετίας είπατε ότι τα επεξεργάζεστε. Τώρα έρχεστε και μας ενημερώνετε και μας τίθετε ενώπιν της διλήμματος να πούμε ναι ή όχι. Προτάσεις για αλλαγές δεν μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε μόνο να πούμε ναι ή όχι. Και εφόσον μας μεταχειρίζεστε έτσι, στο κάτω της γραφής το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτη. Δεν είναι μόνο του το Συμβούλιο και η Κομισιόν. Γιατί δεν συμμετέχουμε νωρίτερα. Συζητούμε δύο χρόνια την διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη, κάτι το οποίο δεν ήταν και εύκολη υπόθεση, όπω θα σα πούν και οι δύο συγγητέ, και τώρα απλώ διευρύνεται. Μερικέ διευρύνσει μου φαίνονται καλέ, αλλά γιατί μα ενημερώνετε τώρα μόλι για αυτέ. Και ιδίω εάν κάτι δεν μου φαίνεται καλό, πάλι δεν μπορώ παρά να πω μόνο ναι ή όχι. Μα δεν μπορεί αυτό να είναι το μέλλον μα. Και πώ πώς το βλέπετε αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν εμπλέκεται το Κοινοβούλιο ενωρίτερα. Γιατί αποκλείεται στην πράξη το Κοινοβούλιο παρόλο που συναποτελεί μέρος του νομοθετικού σώματος στην Ευρώπη. Και είναι απαραίτητη συμβολή του για την υλοποίηση των έργων αυτών. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Η κυρία Γιάννα μόνο ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, Να πω κάτι στον Μίκαελ για το ελεγκτικό συνέδριο σε σχέση με τους λιμένες και τους αερολιμένες. Δεν μας έχει πείσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλές φορές η κριτική η οποία έγινε είναι κάτι το οποίο ήρθε στην επικαιρότητα στην κορυφή της οικονομικής κρίσης. και νομίζω ότι και σε μικρή κλίμακα θα πρέπει να υπάρξουν ε, ε, το δυνατότητες ε, βοήθησης γιατί νομίζω ότι το να επιδιώκει κανείς μόνο τους πολύ μεγάλους λιμένες και τις πάρα πολύ μεγάλες λιμενικές εγκαταστάσεις και μεγάλα σκάφη κτλ είναι κάτι το οποίο δεν είναι από μόνο του σωστό. Νομίζω ότι θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι έχουμε μία πυκνότητα μικρότερων υποδομών η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί και δεν θα πρέπει να αγνοούμε τον τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφωθεί ακριβώς η κατάσταση στην Ελλάδα. Συμφωνώ μαζί σου Μιχαήλ. Αλλά σε σχέση με το ελεγκτικό συνέδριο νομίζω ότι τα πράγματα ίσως να είναι και τελικά κάπως περισσότερο περίπλοκα. Πάλι ο κύριος Κράμερ. Είχα ξεχάσει να πω πριν κάτι. Οι τσεχικοί σιδηρόδρομοι πρότειναν ε, στους γερμανικούς σιδηροδρόμους να στείλουν μία ταχύα από την ε, Πράγα, από το στο Πασάο στο Μόναχο. Μένει 1,1 χιλιόμετρο κενό. Μήπως εκεί μπορεί να υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα 1,1 1100 μέτρα μένουν και θα έχετε μια θαυμάσια σύνδεση μεταξύ Πράγας και Μονάχου. Με ταχεία, με ταχύ τρένο. Ακολουθεί τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Βερσίνη. Δεν σας μένει πολύς χρόνος, αλλά ε, από σας περιμένουμε απαντήσεις. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι ορισμένες ερωτήσεις ίσως ξεφεύγουν από την αρμοδιότητά σας. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο συνεκτικός ε, και ακριβής απαντήσει μου αρχικά για να απαντήσω στον κύριο Έρτσουκ. Η αναθεώρηση των κατευθύνων γραμμών TNT ε, ε, είχε προβλεφθεί στον ίδιο το κανονισμό ξεκινώντας από το 2023. Σε αυτή τη φάση δεν προβλέπεται ε, να εγκινηθεί μία αναθεώρηση του, του κανονισμού TEN-T. Και μπορεί να σας φαίνεται μακρινή αυτή η ημερομηνία. Και αυτό όμως συμβαίνει επειδή κατά την υιοθέτηση του κανονισμού οι συνομοθέτες θεώρησαν ότι για να θεσπιστεί ένα ε, πραγματικό διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών πρέπει να προβλέψουμε μια σταθερότητα και προβλεψιμότητα για όλα τα διαφορετικά μέρη. Ε, γι' αυτό και με τις σημερινές κατευθυντές πράξεις θέλουμε να δείξουμε πώς ε, αυτοί οι χάρτες ε, και ο κανονισμός μπορούν να ε, ακολουθούν πιστά τις προβλέψεις του δικτύου και τι ανάγκε του δικτύου, ε, λαμβάνοντα υπόψη και την πρόοδο που έχει σημειωθεί, χωρίς να αλλάξουμε όμως την σφαιρική μας στρατηγική. όπως αυτή είχε διαμορφωθεί το 2013 και προβλέπει το, ένα πλαίσιο μέχρι το 2023 τουλάχιστον. Προς απάντηση του κυρίου Βαντερκάμπ και του κυρίου Κράμερ, μας ρώτησαν ποια είναι η σύνδεση με τη χρηματοδότηση. Στην ουσία αυτό το εγχείρημα που είναι τεχνικό εγχείρημα για να αναδείξουμε ακριβώς την πραγματικότητα στο δίκτυο ε, δεν συνδέεται με την ε, χρηματοδοτική αρρωγή προς τα ίδια τα έργα. Αυτά διέπονται στον κανονισμό για τον μηχανισμό διασύνδεσης στην Ευρώπη. Γι' αυτό και η επαλήθευση της προσθέμενης ευρωπαϊκής αξίας που ανταποκρίνεται σε ένα σύνολο κριτηρίων που έχουν οριστεί σε αυτόν τον κανονισμό μας επηρεάζουν εδώ. Και σε αυτό το πλαίσιο θα εφαρμόσουμε τις ε, συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου. Έχουμε πολυάριθμες ε, εκθέσεις που έχουν υιοθετηθεί από το Ελληνικό Συνέδριο για την χρηστή διαχείριση των ευρωπαϊκών ε, πόρων στο σύνολό τους, όχι μόνο για τον μηχανισμό διασύνδεσης στην Ευρώπη, ε, για να δίνουμε μια κατά το δυνατόν αποτελεσματική ε, στήριξη με βάση τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Δεν θέλουμε ε, να έχουμε μια κατακαιρματισμένη εικόνα, θέλουμε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό αποτέλεσμα. Ένα άλλο στοιχείο απάντησης, τα μεγάλα έναντι των μικρών έργων. Μπορεί στο παρελθόν όντως η έμφαση να δινόταν στα πολύ μεγάλα έργα. Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξετάσει και τα πιο μικρά έργα, ιδίως διασυνοριακά, στον διαγωνισμό για τον μηχανισμό διασύνδεσης που τρέχει αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ε, συγκεκριμένος ορισμός ότι αφορά τα μικρά έργα τύπου αυτού που αναφέρατε, τη διασύνδεση με τη Γερμανία. Πιο μικρά έργα λοιπόν, σιδηροδρομικά που μπορούν να μας δώσουν καλύτερη συνδεσιμότητα στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τις ε, αξιολογήσεις περιβαλλοντικού αντικτύπου, είναι μια απέτηση του κανονισμού για το μηχανισμό διασύνδεσης στην Ευρώπη και συστηματικά ε, ελέγχεται κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις του ενωσιακού δικαίου σε ό,τι αφορά την ε, ανάλυση περιβαλλοντικού αντικτύπου. Τώρα για τις ερωτήσεις που αφορούν πιο συγκεκριμένα έργα. Απαντώ στην κυρία Γιάλα Σάντερς. Σύνδεση Βαγιαδολίδη μεταξύ Σανταντέρ και Βαγιαδολίδη Βικτόρια από την άλλη. Ουσιαστικά, εδώ πρόκειται και το ψήφισμα που υιοθετήσαμε για τους χάρτες, γιατί αυτές οι δύο γραμμές παραμένουν μεικτέ γραμμέ, δηλαδή μπορούν να περάσουν στο δίκτυο υψηλή ταχύτητα. Έχουν αναλάβει αυτή τη δέσμευση οι ισπανικέ αρχές και η εκπροσώπησή του αυτή τη στιγμή, μάλλον η αναπαράστασή τους στου χάρτες ε, δεν αλλάζει σε σχέση με τους προηγούμενους χάρτες. Οι δύο γραμμές, το κόκκινο και το μόβ, ε, ε, αντιστοιχεί στον, ε, στον κάθε τύπο. Το ίδιο ισχύει και για την Αλμερία Γρανάδα. Από την άλλη, αυτή η γραμμή επιβαίνεται ως συμβατική γραμμή του κύριου δικτύου για τον ορίζοντα 2030. Το δίκτυο υψηλής ταχύτητας προβλέπεται για αυτή τη γραμμή, αλλά για αργότερα, μετά το 2030. Γι' αυτό και δεν υπάρχει αυτή αναφορά στον χάρτη αυτή τη στιγμή. Για την κυρία Σενάλοβα. Για το δίκτυο στην Τσεχική Δημοκρατία. Με τα χαράς ε, να το εξετάσουμε και να το συζητήσουμε πιο λεπτομερώς, όμως η καταξιδιώτηση πράξη, ε, την οποία εξετάζουμε σήμερα, δεν ε, επηρεάζει σε καμία περίπτωση το τσεχικό δίκτυο. Δεν υπάρχει κανένα αίτημα ε, τροποποίησης ε, του δικτύου από τις τσεχικέ αρχές. Δεν θα αλλάξει λοιπόν ο χάρτης σε σχέση με το 2013. Να το εξετάσουμε λοιπόν και να το επαληθεύσουμε. Πολύ πιθανό να πρόκειται για το επόμενο, την επόμενη εκδοχή που θα υιοθετήσουμε. να το διευκρινίσουμε. Όμω μπορώ να σα καθισχάσω ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή προ το παρόν και να απαντήσω τέλο στην κυρία Δεμόντε. Ε, για τον ε, διάδρο εμπορματοκινητήων ε, υπαριθμών 11 είναι κάτι το οποίο την χάνει διαπραγμάτευση σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, όμως είναι διαφορετικό και ξεχωριστό από το δίκτυο TNT. Το σύνολο των λιμένων που αναφέρονται αποτελούν τμήμα του ε, δικτύου TNT σήμερα και ε, η λειτουργία τους ε, διέπεται από το πλαίσιο του διαδρόμου Βαλτικής Αδριατικής. Αυτά από μένα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Βερσινή. Θα συνεχίσουμε. κλεισμένο των θυρών. Ευχαριστώ όλους όσοι παρέστησαν ε, μέχρι αυτή τη στιγμή. Τους ε, παρακαλώ όμως να αποχωρήσουν διακριτικά και θα τα ξαναπούμε αύριο. Ευχαριστούμε και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και δημοσιογράφους ε, που ενδέχεται να βρίσκονται στην αίθουσα. Παρακαλώ να αποχωρήσουν.